chers collègues, si vous voulez bien prendre place, je vous... Καθίστε παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, για να αρχίσουμε. Στο σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης θα σας παρουσιάσω το σχέδιο έκθεσης που συνέταξα εγώ βάσει το όσων μου αναθέσατε για ένα σημαντικό ζήτημα. Όχι σημαντικό επειδή ασχολούμαι εγώ, αλλά επειδή πρόκειται για ένα θέμα από το οποίο θα έχουμε δυσκολίες και έχει να κάνει με την ευθύνη του κράτους σημαίου ό,τι αφορά το σεβασμό της οδηγίας 2013 για την εφαρμογή της συμφωνίας που σύμψαν οι ενωσοπιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των εργαζομένων στις μεταφορές. Συμφωνίες ECC-ETF. Ε, Σχετικά με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006 και για την τροπήση της οδηγίας 1999-63. Στο ζήτημα αυτό θα πρέπει να έχουμε κάποια στοιχεία κατά νου. Καταρχήν, ε, κάποια ιστορικά στοιχεία ότι όλη αυτή η συζήτηση Βρισκόμαστε τώρα στο 2012, αλλά όλη αυτή η συζήτηση κατά κάποιο τρόπο ξεκίνησε με αφορμή το ατύχημα του Έρικα το Δεκέμβριο του 1999. γιατί όλοι θα θυμούνται ότι όταν έγινε αυτό το ναυάγιο οι συνθήκες ελέγχου του σκάφους και της πιστοποίησης ε, που είχε γίνει επί του σκάφους πριν ε, κάποιο καιρό και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ε, κατάρτιση του πληρώματος αναφέρθηκε. αναφέρθηκε. Όλα αυτά αναφέρθηκαν και στο διεθνές πλαίσιο έγινε η διαπραγμάτευση της Συμφωνίας για την Αυτική Εργασία το 2006. Δηλαδή 7-6-7 χρόνια μετά. Και σε αυτό το πλαίσιο μια συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων έλαβε χώρα μια συμφωνία η οποία συμπεριλήφθη στην οδηγια 2019 2009-13 που πρέπει τώρα να τα σε εφαρμογή. Έχουμε προβλήματα και επί ε, και επί του περιεχομένου. Λοιπόν, για το περιεχόμενο. Να σας πω ότι η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας ε, περιλαμβάνει μια σειρά διατάξεων που δεν βρίσκονται στο κείμενο που μας παρουσιάζεται μας σήμερα, που μας προτείνεται σήμερα, κυρίως ό,τι αφορά την πιστοποίηση, καθώς η πιστοποίηση αυτή περιλαμβάνει κάποια στοιχεία που σχετίζονται με το μισθό και με τις αρχές η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αρμόδια να ασχολείται με το θέμα του μισθού, έτσι λοιπόν δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια διάταξη. Υπάρχουν ε, κάποια ερωτηματικά σε σχέση με τις προθεσμίες μεταφοράς στο ιστορικό δίκαιο. Τέθηκαν και αυτά τα ζητήματα. Καθώς και ερωτηματικά σε σχέση με τις συνθήκες πρόσληψης ε, του πληρώματος. Αυτή η δυσκολία οδήγησε την ε, Επιτροπή να προτείνει δύο διαφορετικά κείμενα. Ένα κείμενο που εξετάζεται τώρα από την Επιτροπή Μεταφορών και νομίζω ότι ο κύριος Σίμψον είναι εισηγητής. Πρόκειται για ένα κείμενο που ε, αφορά την ευθύνη του κράτους λιμένα και κατά κάποιο τρόπο αποσυνδέει το πρόβλημα, δηλαδή την... η ευθύνη του κράτους λιμένα είναι λιγότερο πολύπλοκη να τεθεί σε εφαρμογή από ε, αυτό που αντιμετωπίζουμε εμεί τώρα. Τώρα, σε σχέση με το ζήτημα που αντιμετωπίζουμε εμείς, προστίθεται εδώ μια δυσκολία. Ότι στο Συμβούλιο, ξαφνικά, τα κράτη-μέλη δεν θέλουν ε, καν να ακούσουν ε, για την οδηγία, την εφαρμοστική οδηγία μιας συμφωνίας κοινωνικών εταίρων. Αυτό είναι το πλαίσιο της πρότασης. Εγώ από την πλευρά μου, σε συνεργασία με την ETF, την Ένωση Εργαζομένων στι Μεταφορέ, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ένωση Εργαζομένων στι Μεταφορέ, ε, έχω αντιγράψει κάποιε από τι διατάξει τη ίδιας τη σύμβαση. Ε, θα φανταζόμαι ότι θα υπάρξει πρόβλημα απέναντι στο Συμβούλιο και απέναντι στην Κομισιόν, που θεωρεί ότι η οικονομική σκοπιά δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Όμως, εγώ ειλικρινά νομίζω ότι πρέπει να γίνει η συζήτηση αυτή. Γιατί διαφορετικά... Αυτό που θεωρώ εγώ ότι είναι ένα από τα κύρια σημεία αυτής της νομοθετικής ε, προσπάθειας ε, θα το παρακάμψουμε. Και θα αναφέρω Δύο παραδείγματα. Το θέμα των επιθεωρήσεων, η φύση των επιθεωρήσεων και τα μισθολογικά. Είναι δύσκολα θέματα, φυσικά τα συζητάμε εδώ συχνά στην Επιτροπή μας, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση όλοι έχουν κατά νου και όλοι έχουν δει πέρα από το πρόβλημα της ΕΡΙΚΑ, ανάθετον το πρόβλημα των προσόντων που έχουν ναυτικοί και των συνδικών εργασίας. Ψήφισαμε ένα κείμενο σχετικά με την κατάρτιση των ναυτικών. Ναι, την έκθεση Κρίστενσεν. Αλλά για μια ακόμη φορά δεν αρκεί να λέμε «Α, θα κάνουμε το τάδε και το δίνα» αν δεν ελέγχουμε ότι όλα αυτά εφαρμόζονται. Λοιπόν, δεν ε, θέλω να μακρηγορήσω περισσότερο. Θα αφήσω στους συναδέλφους το χρόνο να καλύψουν το κείμενο. Σας παρακαλώ να δείτε αν συμφωνείτε μαζί μου στα κυρία σημεία. Θα πρέπει να εργαστούμε μαζί με την νομική υπηρεσία για να δούμε πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε το εμπόδιο αυτό αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια πραγματική δυσκολία εδώ στο να πάρουμε μόνο την πρόταση της Κομισιόν, γιατί αν δείτε το σχέδιο οδηγίας που μας έχει υποβληθεί, δεν περιλαμβάνει παρά πολύ ελαφρές διατάξεις σε σχέση με τον ορισμό του πλοίου, του εφοπλιστή, της αναγκαιότητας ελέγχου συμμόρφωσης και για το θέμα του ποιοι είναι αρμόδιοι να ελέγχουν αυτή τη συμμόρφωση. Και με κάτι τελευταίο που έχει να κάνει με την εξέταση των κατοικιλιών και κατόπιν έχουμε και το θέμα της μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο. Σας κάνω κάποιες προτάσεις πιο φιλόδοξες εκεί. Αυτή είναι η δυσκολία ενώπιον της οποίας βρισκόμαστε. Και καταλαβαίνω ότι υπό αυτές τις συνθήκες εσείς θεωρήσετε ότι θα έπρεπε να ασχοληθώ. Λοιπόν, ξεκινάμε τη συζήτηση. Παρακαλώ. Έχει το λόγο κύριε Oui, Madame la Présidente. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που στη παρουσίασή σας διευρύνετε το φάσμα της πρότασης της Επιτροπής. Εγώ εκλέγομαι σε μια περιοχή που έχει πληγεί από το ατύχημα του Έρικα. Και πραγματικά το τραύμα ήταν πολύ σημαντικό για την περιοχή. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μεγάλη τιμή για μας και για τις προσπάθειες που κάνουμε εδώ αυτή η προσπάθεια πρόληψης που κάνουμε. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω. Όσον αφορά τις ε, σημαίες, όσον αφορά την ε, κυκλοφορία στις θάλασσες, πολλά συμβαίνουν και πολλά βλέπουμε. Και αν αυτή η έκθεση μπορεί να αποτελέσει την ευκαιρία να βελτιωθούν κάποιες πρακτικές ιδιαίτερα όσον αφορά τα πληρώματα, τους ναυτικούς. Αυτό σαφώς θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το υποστηρίξουμε εδώ στην Επιτροπή Απασχόλησης. Το πιο δύσκολο βεβαίως θα είναι το θέμα των αποδοχών των ναυτικών, γιατί εδώ βεβαίως η πρότασή μας είναι πολύ πιο φιλόδοξη από συνήθες προτάσεις στην Ευρώπη. αλλά θα μπορέσουμε τουλάχιστον να το συζητήσουμε το θέμα εδώ στην Επιτροπή. Ε, εν πάση περιπτώσει, προσπαθούμε να ακολουθήσουμε κάποιες κατευθύνσεις που μέχρι τώρα δεν τις είχαμε καθόλου ε, διερευνήσει. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Ποιος άλλος θα ήθελε να πάρει το λόγο. Κύριος Φάμπρα. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, όσον αφορά τις ε, προβλέψεις του Διεθνούς ε, Οργανισμού Εργασίας, Ζητώ συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος, δεν είχα βάλει τα ακουστικά μου. Μπορείτε να ξαναρχίσετε. Ναι, εγώ απλώς έλεγα ότι υπάρχει και οι συμφωνίες και οι προβλέψεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας που προβλέπουν ε, κάποια πράγματα και ελπίζω να έχουν ληφθεί υπόψη. Δεν βλέπω κάποιον άλλον να έχει ζητήσει το λόγο. Θα δώσω λοιπόν τον λόγο στο συνάδελφο Μπακ που είναι ο εισηγητής για την Επιτροπή Μεταφορών, για τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, θα μιλήσω γερμανικά, γιατί προετοίμασα την παρουσίασή μου στα γερμανικά. Έχετε δίκιο ότι είμαι εισηγητής ε, για την Επιτροπή Μεταφορών, για τη γνωμοδότηση Επιτροπής Μεταφορών για το θέμα αυτό και βεβαίως και υποστηρίζω αυτά που μόλις είπατε. Θεωρώ ότι η πρότασή σας ε, πάει προς την σωστή κατεύθυνση. Και στην Επιτροπή Μεταφορών διαπιστώνουμε ότι αυτή είναι η ορθή οδός. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων το αποτέλεσμα είναι θετικό. Και αυτό βεβαίως ισχύει όχι μόνο για αυτό το θέμα, αλλά και για άλλους φακέλους. Θα περιοριστώ εδώ μόνο στα δύο θέματα που αναφέρατε. Ενίσχυση των επιθεωρήσεων και ενίσχυση της εφαρμογής των προβλεπόμενων ε, μέτρων. Το θέμα της κατάρτισης των δεξιοτήτων και προσόντων των πληρωμάτων, το άρθρο 5. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και τα επιχειρήματά σας μπορούμε και εμείς να τα υποστηρίξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν κανείς άλλος δεν θέλει να πάρει το λόγο, πρόκειται για διαδικασία στην Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπέργκα της Επιτροπής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Νομίζω ότι η περίληψή σας είναι εξαιρετικά ορθή. Η σημασία αυτής της πρότασης είναι μεγάλη. Η Επιτροπή τι προσπαθεί να κάνει με την πρόταση αυτή όσον αφορά το κράτος λιμένα και όσον αφορά τις προτάσεις μου. Μας εμείς προσπαθούμε ουσιαστικά να ανταποκριθούμε σε αυτό που ζήτησαν οι κοινωνικοί εταίροι το 2009. Προτείνουμε λοιπόν την υλοποίηση αυτών των ε, μέτρων και θα πρέπει εδώ να συνειδητοποιήσουμε και αυτό είναι εξάλλου και η δυσκολία που αντιμετώπισε η Επιτροπή. Αυτή η κοινωνική συμφωνία έχει πιο περιορισμένο ε, περιεχόμενο καθότι η κοινωνική εταίροι ασχολήθηκαν με κάποιες από τις πτυχές αυτής της ε, συμφωνίας καθότι δεν ασχολήθηκαν με το θέμα των χωρών που, από τις οποίες προέρχονται αυτά τα πληρώματα, ούτε με το θέμα των γραφείων που προσφέρουν αυτά τα πληρώματα και τις υπηρεσίες. Αυτό λοιπόν που εσείς ε, θίξατε εδώ είναι η ενίσχυση της κοινωνικής αυτής συμφωνίας. Και βεβαίως ε, ένα από τα θέματα τα οποία δεν μπορούμε να ενσωματώσουμε γιατί δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το θέμα των αποδοχών. Η συμφωνία που ισχύει εδώ βεβαίως είναι θέματα απασχόλησης όπως ορίζονται από την Ομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέματα ασφάλειας και όπως σας είπε και ο εισηγητής, υπάρχουν σημεία τα οποία δεν μπορούν να συμπεριληφθούν για αυτούς τους λόγους. Αυτό λοιπόν που εδώ είναι σημαντικό είναι η υλοποίηση, η εφαρμογή της ε, Διεθνούς ε, Συμφωνίας, η Οδηγία 2009-13 που συμπεριλαμβάνει αυτή την κοινωνική συμφωνία και είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε τι μπορεί να γίνει με το θέμα των πιστοποιητικών. Με την έννοια ότι υπάρχουν τα πιστοποιητικά ναυσιπλοείας και για τα πλοία με ευρωπαϊκή σημαία, αλλά και για πλοία που έχουν σημαία τρίτων χωρών. Τα πιστοποιητικά αυτά, τα οποία σαφώς και προβλέπουν τις υποχρεώσεις των πλειοκτητών αλλά και των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό ισχύει βεβαίως για τις ε, περιπτώσεις πλοίων με ευρωπαϊκή σημαία. Επαναλαμβάνω ότι η οδηγία 2019-2013 συμπεριλαμβάνει κάποιες από αυτές τις προτάσεις, δεν καλύπτει όμως όλα τα σημεία. Κατά τα άλλα συμφωνούμε μαζί σας, μπορούμε να υποστηρίξουμε τις περισσότερες από τις τροπολογίες αυτού του πρώτου σχεδίου όσον αφορά τις αρμοδιότητες των επιθεωρητών, όσον αφορά τις διαδικασίες για τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν σε ένα πλοίο. Και βεβαίως σκοπός όλης της προσπάθειάς μας, όλης της εργασίας μας είναι να αυξηθεί η ασφάλεια και να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια σε ε, πλοία ευρωπαϊκής σημαίας. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Θα ήθελα να πω στον ε, Ρισάρ Φάμπρ ότι η σύμβαση για την Ευτική εργασία του 2006, γιατί περί αυτής συζητούμε, διαπραγματεύθηκε στα πλαίσια του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Περί αυτής ε, ομιλούμε. Ίσως λοιπόν όταν πάμε στη Γενέβη μπορούμε να συζητήσουμε με αυτούς που είναι αρμόδιοι για την σύμβαση αυτή και να δούμε τι προβλέπεται για την μεταφορά της. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω στην Επιτροπή Μεταφορών συμβαδίζεται με την θέση μας, γιατί αυτό ενισχύει τη θέση του Κοινοβουλίου. Εγώ δεν πρόκειται να υποχωρήσω για το θέμα αυτό. Βλέπω ότι υπάρχουν νομικά θέματα και δυσκολίες, αλλά ακόμα και οι τρίτες χώρες έχουν κάποια επιχειρήματα και γνωρίζω έναν δικαστή στο δικαστήριο ναυτικού δικαίου. Είναι ο Ζων Πιέρ Κότ, γνωστός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και αλλού. Ο Ζων Πιέρ Κότ, λοιπόν, μου λέει ότι δεν του αρέσει όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει ξεχωριστά πρότυπα όσον αφορά το ναυτικό δίκαιο. Καθότι θα πρέπει να διέπει και την Ευρωπαϊκή Ένωση το διεθνές δίκαιο. Αν εμείς αποφασίζουμε να κάνουμε συμπληρωματικά μέτρα και άλλες διατάξεις, αυτό αποδυναμώνει το διεθνές δίκαιο. Και σε αυτή την περίπτωση ουσιαστικά ε, κάνουμε κάτι λιγότερο από το διεθνές δίκαιο. Αν λοιπόν θέλουμε να είναι παραδειγματική η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα το ναυτικό δίκαιο που αφορά την ναυτική εγγραφή, θα πρέπει πραγματικά εδώ να εφαρμοστεί το σύνολο αυτής της σύμβασης. Δεν ξέρω βεβαίως ποια θα είναι η εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν διαπραγματευόταν αυτή η σύμβαση. Φαντάζομαι ότι η διαπραγμάτευση αυτή έγινε πριν αναγνωριστεί αν θέλετε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο αυτό σαν ε, νομικό πρόσωπο. Αλλά αυτό που μας ε, ενδιαφέρει είναι τα πλοία που κυκλοφορούν στις ευρωπαϊκές θάλασσες και οι ναυτικοί που εργάζονται εκεί να έχουν μία αντιμετώπιση ικανοποιητική και βεβαίως να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την υγεία των επιβατών και των εργαζομένων σε αυτά τα πλοία. Όσον αφορά τις τροπολογίες, ποια είναι η προθεσμία 17 Οκτωβρίου, μου φαίνεται πολύ νωρίς. Να βάλουμε κι άλλη μια εβδομάδα. Λοιπόν, ναι, θα είμαστε στο Στρασβούργο 24 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι και θα εξεταστούν οι τροπολογίες στις 6 Δεκεμβρίου. Θα προτείνω βεβαίως συμβιβαστικές ε, τροπολογίες για τις 23 Ιανουαρίου και 24 Ιανουαρίου θα τις ψηφίσουμε θα λάβουμε βέβαια υπόψη μας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Σας προτείνω δύο λεπτά διάλειμμα. Ναι, ναι, Bien, chers collègues, si vous pouvez commencer à prendre place, parce que... Καθίστε παρακαλώ, γιατί μετά θα ξεπεράσουμε το χρόνο.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 Too many things. Too important things today. Well, it's quite, quite challenging, yeah. Bien. Alors voilà. Maintenant... Λοιπόν, νομίζω ότι όλοι έχετε λάβει θέση. Προσπάθησαν σύμβουλοι να τροποποιήσουν ε, τους καταλόγους, έχουν ε, τα μέλη, τις ε, κάρτες. Έχετε όλοι τις κάρτες και τις λίστες ψηφοφορίας να, να, να κάνουμε μια δοκιμή. Μπορείτε να ψηφίσετε ό,τι θέλετε. Άρχεται η ψηφοφορία για τεστ, για δοκιμή. Le Άρχεται η ψηφοφορία. Λειτουργούν όλα τα μηχανήματα. Κυρία Χαρκίν, δεν έχετε την κάρτα σας, όχι. Εγώ έχω τη δική μου. Λοιπόν, ψήφισαν όλοι. Έχουμε 38 ψηφίσαντες προς τη στιγμή, 39 με την κυρία Χάρκιν όλα καλά. Στο σημείο 14. Ένα σχέδιο επιστολή για την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Αίτηση για τη μεταλλουργία Γαλλίσια Μέταλ στην Ισπανία. Σας προτείνω να ψηφίσουμε την επιστολή αυτή. Εγκρίνεται λοιπόν, δεν υπάρχει αντίρρηση. Δεύτερη περίπτωση κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Τμήματο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Πρόκειται για την περίπτωση Πεζό στη Γαλλία. Δεν, ε, δεν νομίζω ότι είναι στην επικαιρότητα, είναι παλιά υπόθεση. Αυτή συμφωνείτε όλοι. Μάλιστα, σημείο 16, κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Τμήματο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση την, ε, σε μια υπόθεση στις κατοχώρες που αποτελεί μέρος της μειοψηφίας ανάσχεσης κατά του Ταμείου. Όλοι συμφωνείτε? 17. Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Εδώ πρόκειται για μια υπόθεση που πρέπει να ψηφίσετε, καθώς είχαμε μια προφορική τροπολογία Πρόκειται για μια περίπτωση στην Σουηδία, επίσης χώρα που ανήκει στη μειοψηφία ανάσχεσης κατά το Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Προφορική τροπολογία έχει να κάνει με την παράγραφο 3. Συμφωνείτε όλοι για αυτή την προφορική τροπολογία η οποία θέλει να διορθώσει την αξιολόγηση της κατάστασης γιατί έλεγε το αρχικό κείμενο καλωσορίζει τη σχετικά ε, ταχεία διαδικασία αξιολόγηση, αλλά δεν ήταν ταχεία διαδικασία αυτό. Έτσι λοιπόν, εγώ σα προτείνω regrets the lengthy evaluation period. Συμφωνείτε όλοι, εγκρίνεται η επιστολή με αυτή την τροποποίηση. Σημείο 18, κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Πρόκειται για μια περίπτωση στις κάτω χώρες. Ε, συμφωνείτε όλοι με την επιστολή αυτή. Συμφωνείτε. Πρόκειται για μια περίπτωση κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση στην Ιρλανδία. Αυτή είναι η επόμενη περίπτωση. Χώρα που επισκεφθήκαμε και δεν υπάρχει συνδικάτο για να συζητήσουμε την εφαρμογή του Ταμείου. Συμφωνείτε όλοι, πολύ ωραία. Ευρωπαϊκό μια Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Εδώ έχουμε μια υποδειγματική περίπτωση γιατί πρόκειται για την κινητοποίηση από τη Γερμανία, υποδειγματική χώρα στο κινητοποίηση του ταμείου αυτή, αλλά είναι αντίθετη. Όλοι συμφωνείτε, ωραία. Τελευταία περίπτωση. Μια υπόθεση που αφορά τη Δανία, χώρα που και αυτή ανήκει στη μειοψηφία ανάσχεσης. Το λέω γιατί κανείς δεν γνωρίζει τι ψηφίζουμε. Και ψηφίζουμε σαν μηχανές, ενώ πρέπει να ψηφίζουμε πιο ξεκάθαρα. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση για μια υπόθεση στη Δανία. Συμφωνείτε όλοι? Ωραία. Λοιπόν, φτάνουμε στο σημείο 22. Με συγχωρείτε. Κάποιος έχει ζητήσει το λόγο, παρακαλώ. αποτελώ με αυτής της Επιτροπής εδώ και 9 χρόνια. Δείχνει ότι τελικά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με καμία από αυτές ε, τις ε, προτάσεις. Και θα ήθελα παρακαλώ πολύ αυτό να αναγραφεί στα πρακτικά. Monsieur, Monsieur ε, d'abord je veux... Καταρχήν, με συγχωρείτε που προφέρω λάθος το όνομά σας. Μέχρι τώρα ποτέ δεν μου είχατε κάνει κάποια παρατήρηση σχετικά με αυτό. Και σε όλες τις συνεδριάσεις των συντονιστών, εγώ με τον ίδιο τρόπο προφέρω το όνομά σα, αλλά αν κάνω λάθος, σα παρακαλώ να με συγχωρήσετε. Και να προβείτε σε μόνιμη κατάρτισή μου. Κατόπιν δεν δέχομαι την ε, πρότασή σας, αν θέλετε αυτή την ανταλλαγή να τη βάλουμε στα πρακτικά, γιατί ψηφίσαμε πάνω από έξι προτάσεις και θα έπρεπε να κάνετε την παρατήρηση αυτή τη στιγμή που συζητήσαμε και έβαλα προς ψηφορία την πρώτη από αυτές τις επιστολές. Αλλά αν θέλετε μπορώ να κάνω μια ψηφορία διαδικασίας και να ζητήσω να ψηφίσουμε το σύνολο των επιστολών και να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Αλλά στην περίπτωση αυτή θα πρότεινα ομαδοποιημένη ψηφοφορία. Υπάρχει πλειοψηφία για να προχωρήσουμε σε ομαδοποιημένη ψηφοφορία ηλεκτρονική μορφή για το σύνολο των επιστολών ή πιστεύετε ότι δεν χρειάζεται και ψηφίσαμε όπως έπρεπε στις κατάλληλες συνθήκες. Ο κύριος Σόρη. Κοιτάξτε, Αυτό που μπορεί κανείς να πει όσον αφορά τη γενική παρατήρηση που ακούστηκε για τη διαδικασία αυτή, ναι, μπορεί αυτό να μπει στα πρακτικά. Εγώ θα υποστήριζα ηλεκτρονική ψηφοφορία γιατί νομίζω ότι θα ήταν ταχύτερη και δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε όλες αυτές τις ομιλίες αλλά θα ήθελα να συμφωνήσω με τα σχόλια του συναδέλφου. Πολύ ωραία, το σημειώνουμε και αυτό στα πρακτικά. Φτάνουμε στο σημείο 22. Ψηφίζουμε την έκθεση Χέντελ για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης. Ε, καταρχήν έχουμε την πρόταση ε, να απορρίψουμε την πρόταση της Κομισιόν από την πλευρά του ΣΥΓΙΤΑ. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ της απόρριψης της πρότασης της Κομισιόν. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Δεν εγκρίνεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση, κυρία ΣΥΓΙΤΑ. όχι. Απορρίπτεται λοιπόν η πρόταση αυτή. Τώρα, για την πρόταση αυτή καθ' αυτή. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26. Ρουντσούλη, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Αποσύρθηκαν. Η 37 δεν είναι παραδεκτή. Πάμε στην 38 της κυρίας Εστρέλη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Κυρία Χαρκίν, θα μου πείτε τι ψηφίζετε. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. 25 υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται. Δεν δουλεύει. Μήπως να δοκιμάσετε κάποιο άλλο μηχάνημα. Λοιπόν, κατόπιν. Τέλος πάντων δεν αλλάζει ψηφοφορία. Λοιπόν, πάμε στο συμβιβασμό D. Άρθρο 16 1. υπέρ. Κατά. Συγγνώμη. 39, 39 Χέντελ. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε στο συμβιβασμό D, δέλτα, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 42. Ζητά να διαγραφεί το άρθρο 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 43. Θέλετε παλήθευση για την 42. Να ψηφίσουμε. Κυρία Χάρκιν, τι ψηφίζετε. Κατά, μάλιστα. Και ο κύριος είναι κατά. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 22 υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44. Μανέσκου. Υπέρ. Να επαληθεύσουμε τη 43. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Υπάρχει μία παραπάνω κάρτα από το ΕΛΚ. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 31 υπέρ, 16 κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στη 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. 21 υπέρ. 16 κατά. Εγκρίνεται. 45 Μανέσκου υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46-47 δεν είναι αποδεκτές. 48. Δεν είναι γλωσσική η τροπολογία. Ωραία, πρέπει να την ψηφίσουμε. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος για 48. Πέρας. 23 υπέρ, 24 κατά. Μπορείπτεται. 50 εστρέλα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51 εστρέλα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται, 53 υπέρ, κατά, αποχές, να δούμε να το ελέγξουμε. Με επαλήθευση της 53 ψήφισατε όλοι. 22 υπέρ, 24 κατά. Απορρίπτεται. 54 του Τόμας Μαν, λέει η πρόεδρος. 54. Τόμας Χέντελ. Τους ακούω ε, φορές να μιλάνε μαζί. Λοιπόν, Τόμας Χέντελ, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 55. Μάλλον επαληθεύσουμε την 54. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 22 υπέρ, 24 κατά, απορρίπτεται 55 ροντζούλη υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 57, το μασέντελ υπέρ. Υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 58, του ιδίου υπέρ. Κατά. Αποχές, νομίζω ότι εγκρίνεται. 59 του ιδίου υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 60 του ιδίου υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 62 του ίδιου υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συνδεσμός Ι, ε, υπέρ. Κατά αποχέ, εγκρίνεται. 66 ροντσούλη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός F. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός G. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 60. Ε, το Τρέλα υπέρ κατά. Και συγκρίνεται. Έχει το μεσχέντελ υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συντά, Συγγνώμη. 71 Εστρέλα υπέρ κατά Ποια εγκρίνεται 72 Εστρέλα υπέρ κατά Εποχέ απορρίπτεται 74 Εστρέλα υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται 75 του συγητή υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται 76 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται 78 Ροντσούλη υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται 79 του ηγητή υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 80 εστρέλα υπέρ, κατά εποχές για να επαληθεύσουμε την 80. το όλοι. Πέρας. 24 κατά απορρίπτεται. Συνδεσμός α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. συμβεσμός Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός Γ σε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συνεχίζουμε για τα εκτιμώντας με την τροπολογία 4 κυρία Στρέλα υπέρ κατά αποχές δεν ξέρουν οι πια τι κάνουν. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5, το μας χέντελ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Καταπέπτει η 6 και περνάμε στην 8 του συγκητή, Υπέρ. Κατά. βοχές, Ρίπτεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 12 του συγητή. Πάλι εδώ διαγραφή του κτήματο 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλήθευση της τροπολογίας 12. Άρχεται ψηφορία. Κυρία Χάρκιν καταψηφίζει. Το δίκαιο Κρίστανσεν Πέρας. 23 υπέρ, 22 κατά. Μία αποχή. Έχετε δίκιο, εγκρίνεται. 14 του είχε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τη 13 μπορούμε να την ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 Θέλετε επαλήθευση? Όχι. 15. Στρέλα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16. Στρέλα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17. Μανέσκου υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18. Του εισηγητή. Για το κτήμα της 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μπορούμε να ψηφίσουμε τώρα Υπεγκρίνεται. Έγραψε απορρίπτεται. Με συγχωρείτε, απορρίπτεται. Μπορούμε να ψηφίσουμε τη 19 της κυρίας Εστρέλα. Υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 Εστρέλα, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 Χέντελ, υπέρ. Κατά, εποχές απορρίπτεται. 22 Εστρέλα, υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται 23 χέντελ υπέρ κατά αποχές αγκρίνεται 24 χέντελ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται λοιπόν να ψηφίσουμε το σύνολο της έκθεσης ηλεκτρονικά άρχεται ψηφορία ο εισηγητής υποστηρίζει την έκθεσή του ψηφίσατε όλοι ηλεκτρονικά Ε, ένας δεν ψήφισε. Ε, ένας δεν ψήφισε. Ένας του ΕΛΚ. Λοιπόν, έλξη ψηφοφορία. 43 υπέρ 2 κατά μία αποχή. Χαίρομαι την εισηγεσία. Τώρα το 23. Έκθεση της κυρίας Μπλινκεβιτσούτε. Έρασμος για όλους και όλες. Στο 1-1 τροπολογία 115 η εισηγήτρια είναι κατά υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός ΙΤΑ, H. Μα Μα αφού είναι σαφές, εσείς δεν βλέπετε, δεν έχετε ο, θέαση του συνόλου από εκεί κάτω. Λοιπόν, συμβιβασμό H υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμό Β υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τις 12 και 119 μαζί είναι ταυτόσιμες υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβιβασμός γεώτα. Πέντε ομάδων υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ζ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 και 130 ταυτόσημες υπέρ κατά χες επαλήθευση για τις 15 και 130 ψήφισαν όλοι έλξη ψηφοφορία 23 υπέρ 22 κατά εγκρίνεται Το 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός λάμδα 5 ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 135 κάστλερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 136 της κυρίας Μπεναράμπ Ατού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός μη 5 ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 Κάστλερ υπέρ κατά αποχές α δεν ξέρω επαλήθευση για την 139 λήθευση Κύριε Κρίστεμψεν, έχετε την κάρτα σας και κύριε Λούντβιξεν επίσης. Ε, ναι, ναι. Έληξε λοιπόν η ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. Η κυρία Χάρκιν ψήφισε υπέρ και άρα 22 έναντι 23 αποχές. Η τροπολογία του κυρίου Κάστλερ όχι, εγκρίνεται. 140 υπέρ κατά πόχες εγκρίνεται 141 μπεναράμ ατού υπέρ κατά πόχες απορρίπτεται επαλήθευση για την 141 Madame Marquine, vous votez le 141 Donc le vote Έληξε 30 υπέρ 16 κατά. Εγκρίνεται. 142 έχει αποσυρθεί. 143. Α, έχει αποσυρθεί και αυτό. Α, μάλιστα. 145 τότε. Ούτε αυτό. Μα δεν μου τα λέτε όλα. 19 και 146 ταυτόσημες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 147 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20 και 148 ταυτόσημες υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 149 της κυρίας Κοστέλο υπέρ κατά χες 150 υπέρ κατά χες επαλήθευση 150 έληξε 41 υπέρ 4 κατά 21 πίπτη, συμβιβασμός νη 5 ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 156 κάστλερ υπέρ κατά ψυχές απορρίπτεται 157 τι επαλήθευση του 156 εντάξει επαλήθευση επαλήθευση επαλήθευση του 156 της 156 Έληξε. Η κυρία Χάρκιν ψηφίζει κατά, 14 κατά 26 λοιπόν, με τρεις αποχάς. Απορρίπτεται πανηγυρικά. 157 Κάστλερ υπέρ. Κατά. Χες απορρίπτεται. Συμβιβασμός πι, υπέρ. Κατά. ΧΕΣ, Εγκρίνεται. 160 Μπεναράμπ Ατού υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 161 υπέρ κατά αποχές νομίζω απορρίπτεται επαλήθευση Madame Marquine Madame Marquine vote pour Κυρία Χάρκιν ψηφίζει υπέρ έληξε 28, 20 υπέρ, 20 κατά, απορρίψτε. Συμβαίνουμε Q, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται 26-165 ταυτόσημες υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνονται άρα 27 και 168 υπέρ, κατά, όχι, δεν 29 και 169 υπέρ, κατά, όχι, εγκρίνονται. 28 και 170 υπέρ, κατά, όχι, εγκρίνονται. 30 και 171 υπέρ, κατά, όχι, εγκρίνονται. 31 και 172 υπέρ, κατά, όχι, εγκρίνονται. 32 της εισηγήτριας υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός ρο υπέρ κατά χε εγκρίνεται. 177 της κυρίας Μπεναράμπ υπέρ κατά απόχέ. εγκρίνεται. 178 υπέρ κατά απόχέ. εγκρίνεται. 33 και 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμό σίγμα 5 ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 34. Η συγκεκριά είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Σύμβασμος ΤΑΦ, πέντε ομάδων υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 35 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 36 και 185 ταυτόσημες υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 37 και 186 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 38 και 188 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 187 κατά πίπτη 189 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 και 190 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός ου 5 ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 και 193 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 42 και 194 ταυτόσημες υπέρ κατά άποχες εγκρινώνται 43 και 195 υπέρ κατά άποχες εγκρίνονται 198 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 199 υπέρ κατά χες εγκρίνεται συμβιβασμό Β. Πέντε μάλλον υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. W υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 46 και 205 ταυτόσημες ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 206 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται απορρίπτεται 47 υπέρ κατά ποχές απορρίπτεται 207 της Μαλίκας Μπεναράμπ υπέρ κατά ποχές απορρίπτεται 48 και 208 ταυτόσημες υπέρ κατά ποχές εγκρίνονται. συμβιβασμός χ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 213 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 214 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 215 της κυρίας Μπεναράμπ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51 και 216 ταυτόσημες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός Y υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 221 υπέρ κατάποχες, εγκρίνεται 53, 54 και 222 υπέρ κατάποχες, εγκρίνονται 224 υπέρ κατάποχες, εγκρίνεται α όχι και 223 και 223 ποιος είναι υπέρ 223 κατά αποχές εγκρίνεται 55 και 225 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 226 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 και 227 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 57 και 229 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 58 και 231 υπέρ κατά βροχές εγκρίνονται 59 και 233 υπέρ κατά βροχές εγκρίνονται 60 και 235 υπέρ κατά βροχές εγκρίνονται συμβιβασμό Ζ υπέρ κατά βροχές εγκρίνεται συμβιβασμός ΑΑ 4 ομάδων υπέρ κατά βροχές εγκρίνεται συμβιβασμός ΒΒ 4 ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. συμβολισμός γάμα γάμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. συμβολισμός δέλτα δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 250 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. συμβολισμός εψιλον ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 και 254 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 68 και 255 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 257 της κυρίας Μπεναράμπ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 260 υπέρ Κατά. Ποιος είπε υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 261 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, Συμβασμό φίφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβασμό GG υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 72 και 266 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 267 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 269 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 268 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται 271 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 και 270 υπερ υπέρ κατά εγκρινόνται. εγκρινώνται 75-272 υπέρ κατά αποχές τα ίδια εγκρινόνται. 274 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 και 273 ταυτόσημες υπέρ κατά ποιες εγκρίνονται 276 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77-275 υπέρ κατά ποιες εγκρίνονται 78 και 277 υπέρ κατά δεν εγκρίνονται 278 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 279 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 280 είναι συμβατή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβασμός ή τα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 και 284 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 81 και 285 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 83 και 287 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 84 και της εισηγητρίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 289 όχι 290 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 291 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά χέρις απορρίπτεται 87 υπέρ κατά χέρ απορρίπτεται 88 υπέρ κατά χέρ ο 90 υπέρ κατά χέρ απορρίπτεται 91 υπέρ κατά χέρ απορρίπτεται συμβιβασμός ε, ε4 ε, τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική γάμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για το 10 του σκεπτικού ή 99 με προφορική τροποποίηση. Υπάρχει καμία αντίρρηση. Αντίρρηση για την προφορική. Όχι. Λοιπόν ψηφίζουμε την 99 όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ κατά αποχές. Πορύπτεται. 3 και 100. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Συμβιβαστική δέλτα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 103 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 104 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτωται. 7 και 106 λέει η ομιλήτρια. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 7 και 107 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Συμβιβασμός φι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός G, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 10 και 113 τα φυτόσημες πολλές ταυτόσημες βλέπω λοιπόν μαζί τις ψηφίζουμε υπέρ κατά εποχές εγκρίνονται το σύνολο τώρα α όχι ξέχασα την 114 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται και τώρα το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικός. Tout le monde a Ψηφίσατε όλοι. 40 υπέρ, μία ψήφος κατά και τέσσερις αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Και τώρα προχωράμε στο 24. Πρόκειται για τη γνωμοδότηση της συναδέλφου Jean Lambert για την ε, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ 2014-2020 κατάρτιση του προγράμματος Δικαιώματα και Ιθαγένεια. Ένα παράγραφος 1. Τροπολογία 33 του Τόμας Χέντελ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δέλτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έψιλον. Ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41. Όχι. Όχι. Όχι. 38. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41. Μινοντόρα κλειβέτη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14. Συγγήτριας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 45. Χέντελ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 46 του ίδιου υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 47, Μάνερ και υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. F, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. G, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 κούντς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τρεις τροπολογίες ταυτόσιμες. Η 1 συγγήτριας, 20 του Χέντελ και 21 της κυρίας Χάρκιν και Μάνερ. Όσον αφορά τον τίτλο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3α. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Β, συμβαστική Β, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα την 24, κούν υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 25 Σίμπελ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 Στάινρου και Σίμπελ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 Ηχηγήτρια υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Σι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 κλειφτή και Άρκινς η 32 υπέρ κατά α όχι καταπίπτουν οι 31 και 32 άρα ψηφίζουμε την 8 της ηγητρίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 της υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο του κειμένου με ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ όλοι ψήφισαν Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. 40 υπέρ, 2 κατά. Συγχαρητήρια, κύριε Συγγήτρια. Σημείο 25 της ημερήσιας διάταξης. Είμαστε στην έκθεση της Βερόνικα Λόπε Φοντανιέ όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλληλεία Πρόκειται για γνωμοδότηση για την Επιτροπή Αλίας. Ο κύριος Καντέκ είναι ο εισηγητής. 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 117. τσούπερ υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται 31 της ηγήτριας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, συγγνώμη, 118 Τσούπερ υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 32 συγγήτριας υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 33 της συγγήτριας υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται γιώτα συμβαστική υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 35 της υπέρ, κατά δεν ψηφίζεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 122 Κρίστενσεν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 συγγήτρια υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. J, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 126, σούπερ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 39, α, ξέχασα το κάπα, κάπα, συμβαστική, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 της ηγήτριας, υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται 127 ζούμπερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 40 εισηγήτρια υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ. Κατά αποχές. 41 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε. Τέλος. Εγκρίνεται. 129. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 140. Υπέρ. Κατά. 42. Υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. Ε, ψηφίζουμε τη 43, την 131 της εισηγήτριας και της κυρίας Λάμπερτ με μια προφορική στη δεύτερη γίνονται ταυτόσιμες αυτές οι δύο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται και οι δύο 142, Κρίστενσεν υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 44 της υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45 της υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46 της υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 48 εισηγήτρια υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51, συγχύτρια, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική λάμδα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53 της υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 144, σούμπερ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 54 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 148 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 152 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 56 συγγήτρια υπέρ 56. 56 συγγήτρια, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 57 της ίδιας, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 58 της ίδιας, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το 146 ψηφίζουμε. Ζητώ συγγνώμη για μια κατάργηση. Στο άρθρο 34, ε, η τροπολογία 146, Ζούμπερ. Επαναλαμβάνω τροπολογία 146 της κυρίας Ζούπερ για την κατάργηση, εξάλληψη του άρθρου 34. Υπέρ, κατά, Αποχές. Η 146 δεν εγκρίνεται. 59 υπέρ της εισηγήτριας. Υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60 της ίδιας υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 61. Συγγήτρια υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62. Της ίδιας υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 156 του κυρίου Κρίστενσεν με προφορική υπέρ Α, συγγνώμη, το 64 πρώτα της ηγήτριας, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 156, με προφορική τροπολογία, δεν υπάρχει αντίθεση, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 65 της ηγήτριας, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 157 Κρίστενσεν, με μία προφορική, ψήφισμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 66 ηγήτριας υπέρ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 Εγκρίνεται 79 με δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα μέχρι small scale fishery. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά. Ποιος είναι υπέρ? Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές. Επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 79. Ψηφίσατε. Τέλος. 21 υπέρ, 15 κατά. Εγκρίνεται. 80, Κρίστενσεν υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 81, Ζούμπερ υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 1, Συγγήτρια υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Α, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Β, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 ζούμπερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Α, συγγνώμη, το 5, το 5. Το 5 της εισηγήτριας υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 88, Κρίστενσεν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 89, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6, εισηγήτριας υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα τη συμβαστική C, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 9 συγγήτριας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 92 με μία προφορική της κυρίας Ζούμπερ υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 10 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 Κρίστιντσεν. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 της κυρίας Σούπερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 εισηγήτρια υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 Κρίστενσεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 σκεπτικό 35 14 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 Κρίστενσεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική ε υπέρ κατά εγκρίνεται 36 υπάρξει τροπολογία 101 σε δύο τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Μέχρι capacity Το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε το 101. Υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα οι δύο λέξεις. Υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 Τσιγήτριας. Υπέρ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 ζούμπερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 39 κυρία Ζούμπερ τροπολογία 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 106 Τροπολογία 106. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 18 της υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 της υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 της ηγήτριας, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 της ίδιας, υπέρ. Κατά. Αποχές. Υπέρ της 21. Συγγνώμη, 22, 22. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 της ηγήτριας, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H. Υπέρ. Κατά. Ποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Τσιγήτριας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26. Τσίδιας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27. Της Τσιγήτριας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 114. Κρίστενσεν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28. Τσιγήτριας. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29 της ηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε συμβαστική μη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. 39 υπέρ. 2 κατά, 3 αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. les et là, ça ne change rien, parce qu'il y a quand même le bébé. Mais par contre, celui-là, il est, il est retiré. Nous en venons au... στην ψηφοφορία ενό σχεδίου γνωμοδότηση προ μια ουσιαστική οικονομική και νομισματική ένωση. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση για την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή. Η συγκεκριμένη είναι η κυρία Τάιση. Για τη σύσταση 1. Είχαμε 10 ίδιες τροπολογίες, ε, η τροπολογία 186, Bauer και Όρη, 188 από την κυρία Ντενούτα Σλαζιόβεσκα, η 189 της κυρίας Χίρς και του κυρίου Μπενιάν αποσύρθηκαν. Ψηφίζουμε λοιπόν ε, την 186 και την 188 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Λοιπόν, πάμε στην 190 του κυρίου Μπενιών, η οποία έχει αποσυρθεί. Επομένως, ψηφίζουμε το συμβασμό R από τρεις ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός S από τρεις ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός TAF ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός U που παρουσιάστηκε από δύο ομάδες υπέρ κατά εποχές να επαληθεύσουμε για τον συμβασμό U. Άρχεται η ψηφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 23 κατά, 21 υπέρ. Εγκρίνει. Δεν εγκρίνεται. Λοιπόν, ψηφίζουμε το συμβασμό V από τρεις ομάδες. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασμός W που κατατέθηκε από τρεις ομάδες. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Για τη σύσταση 1 και πάλι. Οι τροπολογίες 187 και 185 καταπιτούν. Έτσι λοιπόν περνάμε στη ψηφορία της τροπολογίας 191 και της τροπολογίας 192 που είναι ταυτόσιμες για τη σύσταση 2 και αφορούν διαγραφή υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να το επαληθεύσουμε. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. 22 υπέρ, 22 κατά. Απορρίπτεται. Σύσταση 3. Οι τροπολογίες 193 και 194 είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Εποχές. Νομίζω ότι είναι το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά καλύτερα να επαληθεύσουμε. Ψηφίσατε τη Πέρασε ψηφοφορία. 22-22. Απορρίπτεται. Για τη σύσταση 6. Έχουμε μια προφορική τροπολογία της κυρίας Μπάουερ που αφορά τη διογραφή. Έχετε εντρήσεις. Όχι. Είναι κατά ο κύριος Σέρκας, δεν μπορούμε λοιπόν να την ψηφίσουμε για τη σύσταση 6. Σημείο 1, 197, Bauer Όρη. Περ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 198. Έχουμε τους δύο συντάκτες. Υπέρ, κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε την 198. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. 22-22. Δύο αποτέλεσμα. Δεν εγκρίνεται. Τροπολογία 199 οι δύο συντάκτες ε, το ίδιο θέμα υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται για τη σύσταση 6 με 4 προφορική τροπολογία από την κυρία Μπάουερ με το ίδιο αντικείμενο διαγραφής ε, αυτής της παύλα. κυρία Σέρκας έχετε αντίρρηση δεν μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε για συστασία 6 5 έχουμε εδώ πάλι πρόταση διαγραφής υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Σύσταση 6. Τροπολογία 195 του κυρίου Σέρκας υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Σύσταση 6, 196 των κυρίων Κορνέλτσεν Λαμπέρ, Πέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μετά έχουμε το εκτιμώντας α, 115 τροπολογία του κυρίου Σέρκας, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός Β υπέρ κατά Αποχές. εγκρίνεται. Μετά έχουμε την ε, τροπολογία 122 του κ. Σέρκας υπέρ κατά Αποχές. εγκρίνεται. Εκτιμώντας D 124 Μπάουερ. όρη υπέρ κατά Αποχές. απορρίπτεται. Καταψηφίσατε. Λοιπόν, επαλήθευση για την ε, τροπολογία 124. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 17 υπέρ, 25 κατά. Πράγματι απορρίπτεται για το εκτιμώντα D. Δέλτα. Συμβιβασμό C. γάμα Από τέσσερι ομάδε υπέρ κατά αποχέ Εγκρίνεται. Έχουμε την 126 του κυρίου Σέρκας, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, εκτιμώντας ή, 127 του ιδίου, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 128 του ιδίου, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, εκτιμώντας G, συμβασμός δέλτα από τρεις ομάδες, υπέρ, κατά, Εποχές εγκρίνεται. Να επαληθεύσουμε το συμβασμό D, δέλτα. Αρχίζει η ψηφορία. Συμβασμός D. Υποστηρίζεται από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες φιλελεύθερους και τους πρασίνους. Πέρας. 25 υπέρ, 19 Κατά. Εγκρίνεται. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ψηφίσουμε... Όταν φτάσουμε στην 135, εγώ θέλω να την αποσύρω την τροπολογία αυτή. Ε, Μάλιστα, ευχαριστούμε. Ούτω ή άλλω όμω δεν θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε την 135 γιατί καλυπτόταν από την ψηφοφορία του συμβιβασμού D. Σας ευχαριστώ όμω για τη διευκρίνηση αυτή. Στο εκτιμώντα G ψηφίζουμε το συμβιβασμό E. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. 25 υπέρ, 18 κατά. Μία αποχή. Εγκρίνεται. Περνάμε στο Εκτιμώντας AIDS, τροπολογία 137 τον κύριο Μπαουρόρη ζητάνε να διαγραφεί. Το εκτιμώντας υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μπορούμε να ψηφίσουμε τώρα το συμβασμό F, που στηρίζεται από τρεις ομάδες, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εκτιμώντας... ΑΗ 142 τροπολογία έρκας περ κατά εποχές εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 143 της κυρίας Χίρς υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Και η τροπολογία αυτή υποστηρίξεται από τους κυρίους Μπενιών και Χάρκιν. Λοιπόν, και πάλι για το I, 144 του κυρίου Σέρκας, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εκτιμώντας J145 τροπολογία, Κορνέλισον Λάμπερτ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά, εκτιμώντας K146 Σέρκας, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Για τον τίτλο 2, τροπολογία 182, πρόκειται για διαγραφή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται για το εκτιμώντα L τροπολογία 147 με του συντάκτε με δύο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται εκτιμώντας M 148 με δύο αντικείμενο και δύο συντάκτε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Εκτιμώντα M Συμβασμός G από τρει ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 150, Bauer Ori. Επιζητεί τη διαγραφή υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έχουμε τώρα το συμβασμό H που παρουσιάζεται από τέσσερι ομάδε. Για το εκτιμώντας 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Για το τίτλο 3, τροπολογία 183, Bauer Ori. Επιζητά την ε, διαγραφή υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Εκτιμώντας O, ε, συμβασμός I ε, από τρεις ομάδες εγκρίνεται. Λοιπόν, εκτιμώντας P, συμβασμός J που παρουσιάζεται από τέσσερις ομάδες, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πηγαίνουμε τώρα στο εκτιμώντα Q. Τροπολογία 98 της κυρίας πιστά τη διαγραφή, υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε το συμβασμό και από τέσσερι ομάδε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά το εκτιμώντας, το το συμβασμό L, από τέσσερι ομάδε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Για το εκτιμώντας R έχουμε δύο τροπολογίες για τη διαγραφή. Η μία από Μπάουρ και Όρη για την, είναι 161 και έχουμε και την τροπολογία 162 που καταδίθηκε από την κυρία Χίρς, υπέρ αυτών των δύο, 161 και 162. Κατά, αποχές, να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για τις τροπολογίες 161 και 162. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 22-22. Απορρίπτεται. Εκτιμώντας S, ε, συνδεσμός M από δύο ομάδες υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. τίτλο 4, τροπολογία 184, Bauer Ori, επιστατή διαγραφή, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Εκτιμώντας ε, τι, 166, για υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εκτιμώντας τι, συμβασμός 1, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εγκρίνεται, με συγχωρείτε. Περνάμε στο συμβασμό O από ως ομάδες υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός πί, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εκτιμώντας W, συμβασμός Q από τέσσερις ομάδες. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και για το εκτιμώντας X, τελευταία τροπολογία 181. Μπάουερ όρη, επιζητά τη διαγραφή του εκτιμώντας αυτού, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 27 υπέρ, 16 κατά και μία αποχή. Σας ευχαριστώ για αυτή την ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ και για αυτά τα μερικά χειροκροτήματα. Αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την ποιότητα της δουλειάς μας. Μας επιτρέπει να καταλήξουμε σε μια χρήσιμη γνωμοδότηση σε κάποιες συνδικές εργασίες δύσκολες. Φτάνουμε στην τελευταία ψηφοφορία για σήμερα το πρωί. Δηλαδή, της έκθεσης Λίτσια Ροντζούλη. Εντροποποίηση οδηγία 2005 για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρηση για την εσωτερική αγορά. είναι γνωμοδότηση προς την Επιτροπή ΙΜΚΟ όπου η συγκήτρια επί της ουσίας είναι η κυρία Μπερναντέτ Βερνιό. 51-52 ταυτόσημες. Κατά αποχές εγκρίνονται. 55 του Μπεναμία υπέρ κατά χες απορρίπτεται. 53 της Νάντιας Χίρς υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Πώς για το 53 όμως παρακαλώ να επαναληθεύετε. Ψήφισαν όλοι έληξε 25 υπέρ 19 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν 55, 56 εννοεί, υπέρ κατά, 56 λοιπόν υπέρ κατά, ποχές εγκρίνεται, 57 υπέρ κατά, ποχές εγκρίνεται, 58 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 59 και 60 ταυτόσημες. Υπέρ, κατά, χες, απορρίπτεται. 6. Επαλήθευση των 59 και 60 άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε 25 υπέρ, 20 κατά. Εγκαρίνονται. Κάτι δεν είχα καταλάβει φαίνεται. Λοιπόν, 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός φι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63, 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 των ιδίων υπέρ κατά υπέρ μάλλον κατά αποχές εγκρίνεται 71 του Θωμά Χέντελ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ήττα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 10 και 74 του Μπαχ και της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική γιώτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 του Θωμά Χέντελ για διαγραφή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 της ηγητρίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 του Θωμά Χέντελ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 της ηγητρίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 του Θωμά Χέντελ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική κάπα K4 πέντε ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85 Χρίστενσεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 Χρίστενσεν διαγραφής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 Μπεναμίας υπέρ ε, Συμβιβαστική λάμδα 5 ομάδων υπέρ κατά 6 ομάδων αποχές Εγκρίνεται 92 Χρίστενσεν υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 93 του Θωμά Χέντελ υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 94 του Θωμά Μάν υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 95 του Μπεναμία και Μπουλάν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 των ιδίων για διαγραφή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 97 Χρίστενσεν και Λούντβιγκσον για διαγραφή υπέρ κατά αποχές ποιος είπε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 της Νάντιας Χίρς και 99 της Ελισάβετ Μορέν Σαρτιέ και 100 του Μπεναμί και 101 του Τζάμπα Όρη και 102 του Μπουλάν και 103 της Γιασλοβιέτσκα. Είναι όλες ταυτόσιμες για διαγραφή. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά ποχές. Οι έξι αυτές τροπολογίες εγκρίνονται και διαγράφεται λοιπόν αυτό το σημείο. 104 της υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 106 του Μπεναμία και Μπουλάν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 107 Ροντζούλη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 108 Χρίστενσεν και Λούντβιγκσον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 109 του Θωμά Χέντελ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 110 καταπίπτει γιατί ενεκρίθηκε 108. 111 Χρίστενσεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 113 του Θωμά Χέντελ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 114 του Θωμά Μαν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 115 Χρίστενσεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 116 ε, ταυτόσημες και 117. Η Χέντελ και Ροντζούλη υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 118 Χρίστενσεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 Θωμαμάν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 Τουρούνεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 Θωμαμάν υπέρ είναι για διαγραφή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 122 Θωμαμάν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τώρα οι ίδιοι με πριν 123, 124, 125, 126, 127, 128 για διαγραφή. Ψηφίζουμε υπέρ κατάποχες. Οι έξι αυτές τροπολογίες εγκρίνονται. 129 του Θωμάμαν υπέρ κατάποχες εγκρίνεται. Συμβιβαστική μη τεσσάρων ομάδων υπέρ κατάποχες εγκρίνεται. Συμβιβαστική κ δύο ομάδων υπέρ κατάποχες εγκρίνεται. 137 της Μαριάν Χάρκιν, που Μαριάν Χάρκιν, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 139 για Σλοβιέτσκα υπέρ κατά αποχές επαλήθευση. Γιατί έχει καιρό που δεν χρησιμοποιήσαμε τα μηχανήματα. 18 υπέρ 24 κατά 2 αποχές. Η 139 απορρίπτεται. 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 της γήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 144 και 145 ταυτόσημες υπέρ κατά Χες εγκρίνονται. 146 τούρουνεν υπέρ κατά χες απορρίπτεται. 147 υπέρ κατά ποιος είπε υπέρ ξανά κατά αποχές εγκρίνεται. 148 χάρκιν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 150 υπέρ της ίδιας κατά αποχές εγκρίνεται. 151 του Θωμά Χέντελ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 152 του ίδιου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 153 του Μπαχ απορρίπτεται. Συμβιβαστική νη 6 ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Et nous mettons en voie le compromis Συμβαστική όμικρον. Υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 164 χάρκιν υπέρ κατά. Ποιος είπε παιδιά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Α, καλά, επαλήθευση, επαλήθεύση, επαλήθευση 164. Ψηφίσατε όλοι και όλες ελειψε Υπέρ 30, 15 κατά καμία αποχή εγκρίνεται πανηγυρικά. Ψηφίζουν λοιπόν τώρα την 166 και 167 που είναι ταυτόσιμες του Ρούνιν και Χίρς υπέρ, κατά, ποιε εγκρίνονται. 168 και 169 των ιδίων υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 170 είναι συμβατή υπέρ κατά χες εγκρίνεται 171 Thomas Χέντελ Paul Murphy, υπέρ κατά ποχές εγκρίνεται 173 Χέντελ Murphy και 175 Harkin, υπέρ κατά χες εγκρίνεται 177 Christensen, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 178 Χάρκιν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 179 Χάρκιν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 Είμαστε στο σκεπτικό τώρα. 18 υπέρ κατά χες εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά χες απορρίπτεται. 20. Α, ψηφίσαμε, ψήφισαμε. Ψηφίσαμε. Το 19 τώρα την 20. Υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 21. Υπέρ, κατά Χες. εγκρίνεται. Συμβιβαστική α υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική β υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. 32 του Τζάμπα ο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 της εισηγητρίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 της εισηγητρίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική γάμα τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 ανάδεια χείρς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική δέλτα πέντε ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελευταία μας ψηφοφορία ηλεκτρονικά για το σύνολο. Άρχεται. Ψήφισαν όλοι και όλες έληξε 40 υπέρ 2 κατά 3 σαποχές συγχαίρουμε την κυρία Ραντζόλη Με. Παρακαλώ του σοσιαλιστέ και σοσιαλίστριες Κύριε Σάρκα Κύριε Σέρκα είναι πολύ προβληματικό γιατί πήγαμε γρήγορα και ο σκιώδης εισηγητής για το επόμενο δεν έχει έρθει ακόμα. Τι να κάνουμε τώρα. Κύριε Πριότε, τι μπορούμε να κάνουμε. Θέλετε να τον περιμένουμε, μπορείτε να τον φωνάξετε. Τι να κάνουμε. Να αρχίσουμε, μάλιστα. Λοιπόν, θα εξετάσουμε λοιπόν τώρα το 28 που θα δώσουμε πρώτα το λόγο στην εισηγήτρια Νάντια Χίρς. Ησυχία παρακαλώ. Ησυχία την έκθεσή της, την έκθεση πρωτοβουλίας της, το σχέδιο έκθεσης πρωτοβουλίας της για τη μεταχείριση των μεταναστών κλπ. Για αυτή την έκθεση έχουμε ενισχυμένη συνεργασία με την Επιτροπή ΕΛΕΦ όπου η συγητής θα είναι ο Φίλιππος Κλάες των μη εγγεγραμμένων. Δίνω λοιπόν το λόγο στη δική μας εισηγήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση βασίζεται σε μια μελέτη της Επιτροπής και σε διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις. Προσπάθησα λοιπόν εγώ να συμπεριλάβω όλα αυτά σε μία έκθεση. Πρέπει όμως να σας πω ότι μόνο τα κεντρικά σημεία αυτών των παρουσιάσεων ενσωματώθηκαν. Γι' αυτό και από τις τροπολογίες σίγουρα θα συμπληρωθεί το κείμενό μου. Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να εξετάσουμε τα βασικά σημεία. Θα πρέπει να δούμε πώς έχει η δημοκρατική εξέλιξη στις χώρες μας, οι αδυναμίες και οι ελλείψεις στην αγορά εργασίας και οι αδυναμίες και ελλείψεις ε, που μπορεί να καλυφθούν από τους μετανάστες στις αγορές εργασίας. Πρόκειται για άτομα που έρχονται από τρίτες χώρες. Χρειαζόμαστε άτομα βεβαίως με προσόντα και δεξιότητες. Πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλίας όπως είπατε. Και αυτή η πρότασή μου περιέχει μια νέα ιδέα. Μια νέα ιδέα που είναι η δημιουργία ενός ε, συστήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προσέλκυση και την ενσωμάτωση μεταναστών οι οποίοι έχουν κάποια κατάρτιση και κάποιες δεξιότητες. Αυτό βεβαίως ε, γνωρίζοντας ότι το θέμα της μετανάστευσης είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Παρόλα αυτά θέλουμε να δούμε αν ένα σύστημα προαιρετικό μπορεί να δημιουργηθεί όπου σε εθελοντική βάση και κατά περίπτωση θα επιλέγουν τα κράτη-μέλη αν θέλουν να ενσωματώσουν, αν χρειάζεται να ενσωματώσουν κάποιους μετανάστες. Από τη μία μεριά λοιπόν έχουμε όλα αυτά τα άτομα που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ενσωματωθούν, να μάθουν τη γλώσσα των χωρών στις οποίες θέλουν να εγκατασταθούν και αυτό βεβαίως να γίνεται με τις καλύτερες συνθήκες. Από την άλλη μεριά το θέμα της αφομοίωσης. Δεν θέλουμε να υπάρξει αφομοίωση, θέλουμε οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να κρατήσουν την ταυτότητά τους. Βεβαίω, εδώ οι διάφορες χώρες έχουν διαφορετική παράδοση και γι' αυτό και πιστεύω ότι θα υπάρξει έντονη συζήτηση σε εθνικό επίπεδο. Κάνουμε λοιπόν εδώ κάποιες προτάσεις και θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε στους μετανάστες τη δυνατότητα να μάθουν τη γλώσσα των χωρών στις οποίες θέλουν να εγκατασταθούν, έτσι ώστε να μπορέσουν να ενσωματωθούν. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει καν αυτή η δυνατότητα για αυτούς. Δεν τους προσφέρεται η δυνατότητα. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω είναι οι φοιτητέ. Όλοι αυτοί δηλαδή οι οποίοι σπούδασαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους οποίους δεν υπάρχουν οι βέλτιστες συνθήκες έτσι ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν και να εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι ανόητο κατά την άποψή μου, καθότι επενδύουμε σε αυτούς τους ανθρώπους όσο σπουδάζουν. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια χρόνια και να εργαστούν. Αλλά θα πρέπει να τους αφήσουμε τη δυνατότητα να επιλέξουν αφού σπούδασαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν το επιθυμούν, να μπορέσουν να έχουν και μια επαγγελματική εμπειρία, δραστηριότητα στη χώρα που σπούδασαν. Το άλλο θέμα βεβαίως είναι οι πρόσφυγες, οι οποίοι έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω πολιτικών συνθήκων για πολιτικούς λόγους και οι οποίοι θα πρέπει και αυτοί υπό κάποιες συνθήκες να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού προηγουμένως βεβαίως ε, γίνουν κάποιοι έλεγχοι και κάποια ενσωμάτωση. Η ενσωμάτωση εδώ θα πρέπει να γίνεται βεβαίως το συντομότερο δυνατόν και με συγκεκριμένες συνθήκες. Η ενσωμάτωση αυτών των ε, μεταναστών θα πρέπει εδώ βεβαίως να αντιμετωπιστεί με μια πιο συνολική προσέγγιση και θα πρέπει να βρούμε κάποιες συνθήκες οι οποίες να ισχύουν για όλους και για όλες τις χώρες, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζεται ατομικά η ε, περίπτωση αυτή. Και νομίζω ότι το θέμα βεβαίως της καταπολέμησης των διακρίσεων είναι όλα αυτά θέματα που πρέπει να απασχολήσουν την Επιτροπή. Κάτι άλλο που έχω συμπεριλάβει στην έκθεσή μου είναι το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης. Εδώ βεβαίως υπάρχουν πολλές διμερείς συμφωνίες και συνεννοήσεις, αλλά και για αυτό το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης πιστεύω ότι θα πρέπει να βρεθεί μια πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση. Βεβαίως όλα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά τουλάχιστον να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια και σαφήνεια, έτσι ώστε αυτοί οι οποίοι θέλουν να ενσωματωθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην αγορά εργασίας να έχουν κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες για την κοινωνική τους ασφάλιση, όπως έχουν εξάλλου και οι Ευρωπαίοι πολίτες οι οποίοι εργάζονται σε μια τρίτη χώρα. Σήμερα αυτό δεν είναι δυνατόν να ρυθμιστεί βεβαίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα άλλο θέμα είναι οι λαθρομετανάστες, άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς ε, χαρτιά, οι οποίοι όμως εργάζονται στις χώρες μας. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να νομιμοποιηθούν. Πολλοί από αυτούς βρίσκονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονται παρόλα αυτά, στηρίζουν τα συστήματά μας, είτε πρόκειται λοιπόν για ανθρώπους που εργάζονται στο τομέα της γεωργίας ή στις ε, πόλεις, θα πρέπει να βρούμε ένα σύστημα να τους ενσωματώσουμε και να τους νομιμοποιήσουμε. Επαναλαμβάνω ότι είμαι ανοιχτή σε κάθε συζήτηση και ότι θα περιμένω με μεγάλη χαρά και τις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ πολύ. Jean Lambert. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Χίρς ε, για τη δουλειά που έκανε για το θέμα αυτό, γιατί υπάρχουν κάποια πολύ θετικά στοιχεία αν και έχω κάποια προβλήματα, δεν ε, είμαι υπέρ του point system, υπέρ αυτού του συστήματος βαθμολόγησης ε, ε, και είναι ένα ζήτημα αν επιτρέπεται να, να, βρίσκεται ένας μετανάστης βασίνους τέτοιου συστήματος σε μια χώρα. Επίσης, πρέπει να δούμε το θέμα της αναγνώρισης των προσόντων. Αυτό είναι κάτι που γίνεται όλο ένα και πιο σημαντικό ζήτημα και πώς αξιολογούνται και τα προσόντα. Δηλαδή, μιλώ για τους ανθρώπους που ίσως δεν έχουν τυπικά προσόντα και πολλή δουλειά έχει γίνει στο παρελθόν. Δυνάμει του προγράμματος Equal είναι χρήσιμη αυτή η δουλειά και νομίζω ότι μπορούμε να βασιστούμε εκεί, στην έκθεση αυτή. Κάτι άλλο που θα ήθελα να αναφέρω στις τροπολογίες ίσως είναι ο ρόλος των εργοδοτών στο όλο ζήτημα της ενσωμάτωσης και ποιες είναι οι ευθύνες τους. Και νομίζω επίσης ένα ζήτημα είναι ε, η σύζυγη κατάρτισης, ε, δηλαδή τι συμβαίνει με τους συζύγους των ανθρώπων αυτών όταν ε, έρχονται εδώ για να δουλέψουν και να μπορούν και αυτοί να εργαστούν. Ε, δεν ε, γίνεται αναφορά το πώς το διαχειρίζεται η Κομισιόν. Εμείς εξακολουθούμε να θεωρούμε αυτό το ζήτημα είναι θέμα ιστορικών υποθέσεων ενώ ουσιαστικά είναι θέμα κοινωνικών υποθέσεων και απασχόλησης. Αυτό πρέπει να ενδυναμωθεί. Η διάσταση αυτή πρέπει να ενδυναμωθεί. Επίσης, κάτι που υπόθηκε για την κοινωνική ασφάλιση δεδομένων των αλλαγών στην ομοθεσία για την ενιαία άδεια, για την μπλε κάρτα και σε άλλους τομείς, αυτή η ανάγκη να μετακινηθούμε από αυτές τις πολλαπλές διμερείς διευθετήσεις ε, καθίσταται πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν το τι λέμε και για την κοινωνική ασφάλιση είναι σημαντικό. Δηλαδή να φέρουμε τα δικαιώματα που έχουν οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν κινούνται διασυνοριακά. Αλλά χρειαζόμαστε ένα πιο πολύπλοκο σύστημα. Σήμερα για τους ανθρώπους που μετακινούνται εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχει και αυτό το θέμα για την κυκλική μετανάστευση και είναι πολύ σημαντικό και υποστηρίζω ολοψήφα όσοι υποθήκαν για ε, τους νόμους μετανάστες. Ε, πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να μείνουν στο επίσημο σύστημα. Πολλές φορές ε, δεν αναγνωρίζουμε πόσο ε, εύκολο είναι να εντοπίσουμε πότε έχει αλλάξει η κατάσταση. Δηλαδή πρέπει να δούμε και τι συμβαίνει με τους ανηλίκους όταν φτάσουν στην ηλικία των 18 ετών. Δεν ε, μπορούσαμε να επεκταθούμε πάρα πολύ, γιατί ήταν μια γνωμοδότηση πρωτοβουλία, ε, αλλά σας ευχαριστώ πολύ και θα συνεργαστούμε επικοδομητικά. η κυρία Μπλίκεν Βιτσιούτε. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χίρς. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και πολύπλοκο όταν ε, μιλάμε για την ε, ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας ε, και για την ένταξη των οικογενειών τους. Είναι ένα πολύ πλοκό ζήτημα γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και το δύσκολο οικονομικό πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε. Και ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε αυτή την ένταξη. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε ένα συμβιβασμό στην έκθεση αυτή, Πώς δηλαδή να τα διατυπώσουμε όλα αυτά με αποδεκτό τρόπο για τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να κατανοήσουν ότι η μετανάσταση είναι απαραίτητη για την οικονομία μας. Ενίοτε λέμε ότι Υπάρχουν ήδη 25 εκατομμύρια άνεργοι στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επομένως εμείς πρέπει να βρούμε την κατάλληλη μέθοδο για να καταδείξουμε την χρησιμότητα που έχουν οι των χωρών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη δημογραφική κατάσταση των χωρών μας Πρέπει να δούμε τι γίνεται με την οικονομική ανάπτυξη των χωρών μας. Αν κάνουμε διάκριση κατά των μεταναστών, ε, μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν αυτές οι διακρίσεις και πώς θα διασφαλίσουμε ότι οι μετανάστες ε, από τις τρίτες χώρες δεν υφίστανται τις ίδιες διακρίσεις και ακόμη χειρότερες διακρίσεις σε σχέση με τους ε, εργαζόμενους μετανάστες που είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ πλοκή κατάσταση και πρέπει να το υπογραμμίζουμε συνεχώς ε, στην έκθεση. Θα πρέπει επίσης να προβλέψουμε μια γενική αρχή για την ένταξη των μεταναστών, είτε πρόκειται για μετανάστες ε, τρίτων χωρών, ε, θα πρέπει γενικά όλες οι χώρες να εφαρμόζουν μια γενική αρχή γιατί αν δεν έχουμε του ίδιου κανόνες και τις ίδιες αρχές, δεν θα μπορούμε να διασφαλίσουμε την καλή ένταξη των μεταναστών. Και δεν θα μπορούμε να λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά αυτό το point system, υποστηρίζω όσα είπε η κυρία Λάμπερτ. Ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε λίγο περισσότερο για να δούμε ποια θα ήταν η προσθέμενη αξία του συστήματος αυτού με τη βαθμολόγηση για την ένταξη των μεταναστών τρίτων χωρών. Εγώ θεωρώ ότι είναι δύσκολο ζήτημα. Στην έκθεσή σας δεν ε, δίνεται επαρκή έμφαση στην ε, στάση που έχουμε απέναντι στις οικογένειες των μεταναστών, είτε μιλάμε για τις συζύγους ή τους συζύγους, είτε μιλάμε για τα παιδιά γιατί και όλοι αυτοί ανήκουν στο ίδιο ζήτημα. Δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε ξεχωριστά. Τα μέλη των οικογενειών, δηλαδή των ε, μεταναστών, δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε ξεχωριστά. Σε ό,τι αφορά τώρα τους λαθρομετανάστες, είναι διτό το πρόβλημα. Θα έπρεπε να εργάζονται νόμιμα, να πληρώνουν φόρους ε, και να ζουν με αξιοπρεπή ζωή αφενός, αλλά αφετέρου πώς προσγειώθηκαν ε, στις χώρες μας, πώς μπόρεσαν να έρθουν στις χώρες μας, τι δεν λειτουργήσε και ποιος είναι υπεύθυνο. Θα πρέπει και αυτό να το δούμε. Ουσιαστικά υποστηρίζω την γνωμοδότησή σας ε, και ελπίζω ότι θα εργαστούμε επικοδομητικά και θα ε, έχουμε μια έκθεση που θα ωφελήσει όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Σουγκουράνου. Ευχαριστώ. Πρέπει να πω ότι η έκθεση της κυρίας Σχίστα πρέπει να καλωσοριστεί ιδιαιτέρως. Γιατί νομίζω ότι το πρόβλημα της μετανάστευσης και της αγοράς εργασίας είναι τα πιο καυτά θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σήμερα σε καθημερινή βάση. Νομίζω ότι η συγγήτρια σωστά ως ε, κύρια, εντόπισε τα κυρία σημεία με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε. Μίλησε για τις δημογραφικές αλλαγές που είναι δραματικές, την έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού σε μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ε, αγοράς εργασίας και τη συνεχή μετακίνηση των εργαζομένων μεταναστών θα έλεγα ότι αλλάζουν τα πράγματα. Και αυτό το πρόβλημα, το μεταναστευτικό, δεν ε, είναι πλέον αποκλειστικά πρόβλημα προσφύγων, αλλά τίνει να είναι όλο ένα και περισσότερο ένα ευρωπαϊκό μεταναστευτικό ζήτημα, εργασιακό. Και θα ανέφερα εδώ ότι έχουμε ε, την μετανάστευση των νέων ε, από μια χώρα όπως η Ισπανία προς χώρες όπως η Γερμανία ή το Εμένο Βασίλειο για να ζήτηση δουλειά. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να τα δούμε αυτά πιο προσωπικά και όπου δει να κάνουμε κάποιες διακρίσεις μεταξύ των Ευρωπαίων μεταναστών και των εργαζομένων μεταναστών ως γενική έννοια. Επίσης θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ε, στο σημείο αυτό η εργασία, μετανάστευση και η πολιτική γειτονία συναντώνται. Και θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι έχουμε κάποιους μετανάστες που έρχονται από τις ανατολικές ε, χώρες εταίρους, δηλαδή από τους ε, Ευρωπαίους γείτονες. αναφέρονται και τα παιδιά των μεταναστών. Θα πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα γιατί έχουμε πάρα πολύ ψηλό ποσοστό σχολικής εγκατάλειψης. Και υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα που σχετίζεται με τις οικογένειες. Δηλαδή τα παιδιά που έχουν εγκαταληφθεί στις χώρες προέλευσης από γονείς που μεταναστεύουν για να αναζητήσουν ε, εργασιακές ευκαιρίες σε χώρες κυρίως όπως η Ιταλία και μέχρι πρόσφατα η Ισπανία. Επίσης, πιστεύω ότι η έμφαση που δίνεται στην γλωσσική εκπαίδευση είναι κάτι ευπρόσδεκτο. Ρίτσιδες, ε, να γίνονται κάποιοι έλεγχοι πρώτης ε, αναχώρησης. Αυτό νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλό για την προοπτική που θα έχουν οι μετανάστες και γενικά θα έλεγα ότι η θετική συνεισφορά που έφεραν ε, οι μετανάστες εργαζόμενοι στην ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά θα πρέπει να τονίσετε ίσως παραπάνω. Γιατί εξακολουθούμε να έχουμε πάρα πολλές προλήψεις ε, σε αυτό το τομέα. Και κυρίως ε, εδώ, σε όσους δεν το πιστεύουν αυτό, θα ήθελα να επικαλεστώ τα επίσημα αριθμητικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο η συνεισφορά των ε, μεταναστών εργαζομένων ε, στο συνολικό ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάνω από 1%. Είμαι κάπως σκεπτικός προς το point system, αυτό το σύστημα της βαθμολόγησης. Φυσικά και αυτό θα μπορούσε να συζητηθεί, να ακουστούν τα επιχειρήματα. Και για το πρόβλημα της ε, κοινωνικής ασφάλισης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω είναι κάτι το οποίο κάποια στιγμή θα έπρεπε να υλοποιηθεί αλλά καθώς αυτή τη στιγμή όλοι αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα και στα 27 κρατημέλη, νομίζω ότι θα ήταν κάπως δύσκολο, δεν θα έλεγα ανέφικτο, αλλά δύσκολο. Να προωθήσουμε την εναρμόνιση και να έχουμε ένα πανευρωπαϊκό σύστημα. Όμως ε, είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη η έκθεση αυτή και νομίζω ότι θα συνεισφέρει τα μάλα και θα μας βοηθήσει στο να επιλύσουμε τις βασικές πτυχές της αγοράς εργασίας ε, των μεταναστών σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ελμαρ Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια θα ήθελα καταρχήν να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε τη συνεισφορά των μεταναστών στις χώρες μας και βεβαίως στα πλαίσια του, Συμφωνίας του Δουβλίνου υπάρχουν πολλές περιοχές της Ευρώπης και πολλές πόλεις, μεγάλες και μικρές, οι οποίες πραγματικά χαρακτηρίζονται σήμερα από την παρουσία και την συνεισφορά των μεταναστών. Σαφώς και λοιπόν υπάρχουν κάποιες πτυχές της έκθεσης που θα πρέπει να εξεταστούν και να εμπλουτιστούν. Το θέμα των φοιτητών. Υπάρχουν πολλοί φοιτητές ε, από τρίτες χώρες οι οποίοι έχουν μεγάλες δυσκολίες για να σπουδάσουν και κατόπιν να παραμείνουν. Πολλές φορές δεν τους δίνονται βίζα, παραδείγματο χάρη. Τους δημιουργούνται μεγάλες δυσκολίες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για φοιτητέ, επαναλαμβάνω, από τρίτες χώρες, οι οποίοι θέλουν να παραμείνουν, να σπουδάσουν ή να κάνουν μεταπτυχιακά, μεταπτυχιακές σπουδές στις χώρες μας. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να δοθεί ιδιαίτερη έμβαση σε αυτό το θέμα και συμφωνώ με αυτό που είπατε για τους ε, παράνομους μετανάστες, οι οποίοι όμως εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να βρούμε μια κοινή αντιμετώπιση, γιατί βλέπουμε ότι τα δικαστήρια αντιμετωπίζουν με τελείως διαφορετικό τρόπο τις περιπτώσεις αυτές. Με μεγάλη χαρά λοιπόν θα συνεργαστώ με την εισηγήτρια για να ε, επεξεργαστούμε κάποιες από τις στοιχές της έκθεσης και να τις συμπληρώσουμε. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Τσέρκας. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την κυρία σε την πρωτοβουλία αυτή. Νομίζω ότι είναι θεμελιώδες το ζήτημα αυτό. Αν έχουμε 25 εκατομμύρια μετανάστες στην Ευρώπη, έχουμε ενώπιόν μας ε, μία επιλογή, δηλαδή αν θα είναι 25 εκατομμύρια προβλήματα ή 25 εκατομμύρια λύσεις. Και αυτό εξαρτάται από την ένταξη, για να δούμε αν ένα πρόβλημα θα μετατραπεί σε ευκαιρία και να δούμε την πραγματικότητα υπό όλες τις διαστάσεις που είναι πολύπλοκες. Πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν αυτή η δουλειά. Εγώ θα αναφερθώ μόνο στις παραγράφους ε, 24 και 28 και γίνεται μία αναφορά σε ένα θέμα που έχει να κάνει με το συντονισμό των συστημάτων κοινωνική ασφάλισης γιατί όπω εσεί πολύ καλά αναφέρεστε την πρόταση ψηφίσματός σας Επίση, σχολιάζεται και την ανακοίνωση Κομισιόν τη 30 Μαρτίου 2012. Συμφωνώ με αυτά που λέτε στις δύο παραγράφους αυτές, αλλά νομίζω ότι θα χρειαζόταν να εξηγήσουμε καλύτερα στους συναδέλφους της Κομισιόν και να επιμένουμε γιατί πρέπει να υποθούν κάποια πράγματα γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα του συντονισμού δεν έχει μόνο να κάνει με την αντιαφεσβήτητη πραγματικότητα ότι οι μετανάστες ε, ε θα παραμείνουν στην Ευρώπη αν ε, δεν ε, διατηρηθεί σε κοινοτικό επίπεδο το θέμα τη διατήρηση των δικαιωμάτων του, τότε όταν επιστρέψουν στη χώρα του όλα αυτά θα χαθούν. Λοιπόν, αν εγώ είμαι Ισπανό και πάω στην Αργεντινή για 10 χρόνια να εργαστώ, ε, θα μετρήσουν αυτή την ε, προϋπηρεσία, αυτή την εργασία αν θέλετε, αλλά όχι σε εσά, γιατί εσείς που είστε Γερμανίδα δεν έχετε διμερή συμφωνία με την Αργεντινή. Έτσι λοιπόν είναι ένα θέμα δικαιωμάτων αυτό για τους ανθρώπους που έρχονται στην Ευρώπη. Πρέπει να λυθεί το θέμα ε, του συντονισμού των συστημάτων, αλλά θα πρέπει να δούμε και πώς θα διατηρήσουμε τα δικαιώματα αυτά για πολίτες που βγαίνουν εκτός Ευρώπης. Αυτά διασφαλίζονται σήμερα από διμερείς συμφωνίες ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει επιλύσει αυτό το ζήτημα σε κοινοτικό επίπεδο. Όταν ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες πηγαίνουν έξω, δεν έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα, ούτε οι πήκοοι της χώρες, ε, όταν έχουν ζήσει σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία, έχουν επιλύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τις πολιτικές χώρες και για τους δικούς μας πολίτες που βγαίνουν εκτός της Ένωσης. Και η ΟΚΕ στις 4 ε, Οκτωβρίου ψήφισε μια πολύ σημαντική γνωμοδότηση, ομόφωνα, και πραγματικά χρησιμοποίησαν ε, πάρα πολλέ τεχνικέ ικανότητε, συνεργάστηκαν οι προγνώμονε και με τι υπηρεσίε τη Κομισιόν και πέρα από το ότι θα σα στείλουμε αυτή την έκθεση για να την έχετε, ε, ίσως θα μπορούσατε να δείτε και τη δυνατότητα να συνεργαστείτε με αυτού του εμπειρογνώμονε. Εγώ θα προσπαθήσω να καταθέσω τροπολογίε όχι να διορθώσω τόσα λέτε, αλλά για να προσθέσω όλη την ποιοτική σημασία που έχει το φαινόμενο του συντονισμού των συστημάτων κοινωνική ασφάλισης και όχι στι ε, κοινότικέ χώρε, όχι στη διασυνορική εργασία στην Ευρώπη που αυτό έχει ήδη επιληθεί, αλλά για του εργαζόμενου που ζουν εκτό Ένωση για του δικού του εργαζομένου που βγαίνουν από την Ένωση και δεν ε, μπορούν να διασφαλίσουν ε, την ε, σεβασμό των δικαιωμάτων του επειδή δεν υπάρχει μερή συμφωνία. Ευχαριστώ. Θέλει κανεί άλλο. Αλλιώ η Νάντια Χίρς. Κανεί. Καμία. Θα δώσω τότε το λόγο και στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τον κύριο Μουρέν. Και είχαμε πει για συντονιστές και συντονίστριες στο τέλος, ε, μην το ξεχνάτε. Τα ακούσαν οι συντονιστές και οι συντονίστριες. Δεν μ' ακούνε, αλλά τέλος πάντων. Θα τους κάνω εγώ να ακούσουν. Λοιπόν, ο κύριος Μωρέν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Κομισιόν χαιρετίζει τις εργασίες αυτές του Κοινοβουλίου και συμμερίζεται την ανάλυση του ως προς τη σημασία που έχει η σωστή αντιμετώπιση των μεταναστών. Το θέμα βέβαια θέτει και πολλά προβλήματα δικαιοδοσιών και καταμερισμού των ευθυνών. Η ανάλυση της έκθεσης συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση ή μεταχείριση των μεταναστών και την ανάληψη δράσεων που στοχεύουν στην πλήρη συμπερίληψή τους στη κοινωνική και πολιτική ζωή των χωρών όπου ζουν και στην πλήρη πρόσβασή τους στην κοινωνική περίθαλψη και την αγορά εργασίας. Οι υπηρεσίες της Κομισιόν θα ήθελαν να εμβαθύνουν την προβληματική αυτή για τη πλήρη συμπερίληψη των μεταναστών στην αγορά εργασίας με βάση τις προτάσεις που έγιναν στις αρχές του χρόνου για την απασχόληση και οι δικές σας συστάσεις θα μας είναι ιδιαίτερα πολύτιμες. Και ορισμένες πτυχές, ιδιαίτερα την διεύρυνση των οργανισμών εξέβρεσης εργασίας μεταναστών θα χρειαστεί κάποια νομική εμπειρογνωμοσύνη. Όσο αφορά τους μετανάστες από τρίτες χώρες, όχι την εσωτερική μετανάστευση, τονίζεται την ανάγκη συνεργασίας και κοινή δράση σε ενωσιακό επίπεδο και συμφωνεί αυτό με μία ανακοίνωση της 30 2η Μαρτίου της Κομισιόν για την εξωτερική διάσταση του συντονισμού της κοινωνικής πολιτικής. Άλλες πτυχές που θα έπρεπε να ξανασυζητηθούν είναι πώς θα εφαρμοστούν στην πράξη τα μέτρα αμοιβαιότητας, δηλαδή των συμφωνιών σύνδεσης με ορισμένες χώρες προέλευσης μεταναστών, η σύναψη κοινωνικών συμφωνιών και οι διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών, μελών και χωρών που διαθέτουν μηχανισμούς τέτοιου συντονισμού όπως οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και καλύτερο συντονισμός βέβαια μεταξύ των χωρών μελών. Όλα αυτά είναι τρόποι που εξετάζει αυτή τη στιγμή η Κομισιόν και τονίζετε και εσείς στην έκθεσή σας. Ορισμένοι βέβαια από αυτούς θέτουν και το θέμα της νομικής βάσης του νομικού υποβάθρου. Για να συνοψίσω λοιπόν θα ήθελα να πω ότι αυτά που προτείνει η έκθεση είναι αρκετά φιλόδοξα και θα μας χρησιμεύσουν και μάς για τα μελλοντικά μέτρα αντιμετώπισης και της μεταχείρισης των μεταναστητών. Ε, πολύ ωραία. Ο, λοιπόν η συγγήτρια έχει ό,τι χρειάζεται τώρα και γι' αυτό θα λάβει και το λόγο για να βγάλει συμπεράσματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για όλες σας τις προτάσεις, για τα σημεία που θίξατε. Ένα πολύ σημαντικό, κεντρικό θα έλεγα σημείο, είναι ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κοινή προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται προς εμάς, θέλουμε να τους καλωσορίσουμε, να τους πούμε «ελάτε, είστε καλοδεχούμενοι». Για μένα αυτό είναι το κεντρικό, το κομβικό σημείο αυτών που άκουσα. Αναγνώριση των ε, δεξιοτήτων, των προσόντων που διαθέτουν τα άτομα αυτά. Στην παράγραφο 13 ήδη έχω αναφέρει κάτι γι' αυτό. Πολλές φορές οι δεξιότητες και τα προσόντα των ανθρώπων αυτών δεν αναγνωρίζονται καν λοιπόν σαν εργοδότη, θα πρέπει εδώ να μπορέσει να επιλέξει άλλο σημείο αυτό για το ποιον θα υποδεχτεί και ποιον όχι. Το θέμα της ενσωμάτωσης, ενσωμάτωσης των συζύγων, των συντρόφων, των παιδιών και εδώ η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και η Επιτροπή Απασχόλησης έχουν κάποια, αν θέλετε, κοινά σημεία, αλλά και κάποιες ξεχωριστές αρμοδιότητες. Εμείς είμαστε, αν θέλετε, πιο ειδικοί σε θέματα απασχόλησης. Η ΛΥΜΠΕ για την πιο γενική αντιμετώπιση. Και γι' αυτό και κάποια από τα σημεία που αφορούν αυτές τις γενικότερες πτυχές, γι' αυτό και δεν τις ε, εξετάζουμε εις βάθος εμείς. Αλλά στο σημείο 13 θα βάλω σίγουρα το θέμα της αναγνώρισης των προσόντων. Ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως. Σε πολλές χώρες υπάρχει μεγάλη ανεργία. Σημαντική ανεργία. Απ' την άλλη, στη στρατηγική για το 2020 θέλουμε να ενσωματώσουμε ομάδες ανθρώπων με καλύτερο τρόπο στην αγορά εργασίας. Γυναίκες, παραδείγματος χάρη, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε αντιπαλότητα και ανταγωνισμό μεταξύ διαφόρων ομάδων, ευάλωτων ομάδων, όπως οι μετανάστες, παραδείγματο χάρη, κατά των γυναικών. Οι τρίτες χώρες, εδώ υπάρχει δυνατότητα να ενσωματώσουμε εργαζόμενους από τις χώρες αυτές και θα πρέπει βεβαίως να δούμε ποιο τρόπο αυτό θα γίνει, γιατί όπως είπατε υπάρχουν και οι διμερείς συμφωνίες. Τέλος, το θέμα της ενσωμάτωσης σε τοπικό επίπεδο, στους Δήμους και τις κοινότητες. Εγώ ξέρω ότι η ενσωμάτωση γίνεται πολλές φορές σε τοπικό επίπεδο. Αυτό εξαρτάται από τις δυνατότητες που υπάρχουν ε, για την υποδοχή των παιδιών, παραδείγματος χάρη στους παιδικούς σταθμούς, τα σχολεία. Και αυτό δεν μπορεί να ρυθμιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει σε τοπικό επίπεδο, επαναλαμβάνω, να υπάρξουν λύσεις και μια θετική αντιμετώπιση για να υπάρξει πραγματική ενσωμάτωση στις κοινωνίες μας. Οι κοινότητες λοιπόν θα πρέπει να έχουν τις δυνατότητες αυτές για να διεκπαιρεώσουν αυτήν την αποστολή. Ο κύριος Σέρκας μίλησε για τη γνωμοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής. Ναι, τη γνωρίζω. Είναι μια πολύ καλή πρόταση και βεβαίως εδώ μπορούμε να συνεργαστούμε αφού υπάρχουν ήδη ειδικοί και εμπειρογνώμενες που έχουν σκεφτεί τα θέματα αυτά. Κάτι άλλο που αναφέρθηκε είναι το θέμα των μεταναστών των παράνομων. Πώς ήρθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Γερμανία Ξέρω ότι κάποιοι που είναι παράνομοι σήμερα ήρθαν με νόμιμο τρόπο παρόλα αυτά. Πρόκειται για άτομα που ήρθαν σαν νέοι φοιτητέ ε, ή για να εργαστούν φοιτητέ και φοιτήτριες οι οποίοι ήρθαν να εργαστούν σε κάποια συγκεκριμένα θέση, οι οποίοι όμως τελικά έγιναν παράνομοι. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα, ακόμα και σε αυτούς που ήρθαν με παράνομο τρόπο, αφού βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ήρθαν με νόμιμο είτε με παράνομο τρόπο, από τη στιγμή που είναι εδώ, έχουν εγκατασταθεί και εργάζονται, να νομιμοποιηθούν. Αλλά βεβαίως κάποιοι οι οποίοι ήρθαν με νόμιμο τρόπο, ακόμα περισσότερους λόγους έχουν να ε, στηριχθούν από εμά. Χαίρομαι ιδιαίτερα για όλες σας τις προτάσεις. Χαίρομαι που θα υποβάλλετε και τροπολογίες και πιστεύω ότι αυτό θα μας οδηγήσει σε μια ακόμα πιο επικοδομητική συζήτηση. Σκοπός μας είναι η ενσωμάτωση, η επιτυχημένη ενσωμάτωση σε όλα τα κράτη-μέλη ε, των ε, μεταναστών. Ευχαριστώ λέει Πάνω σε αυτή λοιπόν τη βάση θα εγκρίνουμε το χρονοδιάγραμμα. Ο, η όρια κατάρριξη τροπολογιών λήγει στις 6 Νοεμβρίου και μετά τις τροπολογίες 28-29 Νοεμβρίου. Συμβιβαστικές στις 23 και τελική ψηφοφορία στις 24. Τώρα ίσως να σας εκπλήξει, αλλά επειδή μπαίνουμε στην τελευταία φάση των εργασιών μας, δεν πρέπει να στοχίσουμε στο χρονοδιάγραμμα, αλλιώς θα ζημιώσουμε τους άλλους συναδέλφους που βασίζονται τα δικά μας για να συνεχίσουν και τη, αυτή τη δική τους δουλειά. Μπορεί να είναι τεχνικό θέμα, αλλά απαραίτητο. τελειώσαμε με την κανονική μας ημερήσια διάταξη για το πρωί. Όχι, όχι, πώς όχι. Να με συγχωρεί ο εισηγητής Τζάμπα Σόγκορ, πρέπει και αυτός να μας παρουσιάσει την σχέδιο έκθεσής του για τις ευρωπαϊκές δημογραφικές στα Αυτό θα είναι το τελευταίο σημείο. Έχετε το λόγο. Θα μιλήσω ουγγουρικά. Θα ήθελα να εκφράσω τις ανησυχίες μου καθότι υπάρχουν εδώ πάρα πολύ σοβαρές και αρνητικές ε, συνέπειες ε, αυτής της πρότασης της ε, Επιτροπής. Υπάρχουν εδώ προβλήματα και αντικρώμενα συμφέροντα θα έλεγα με πολλές χώρες. Και πραγματικά θα υπάρξουν και πολύ σοβαρές πολιτικές συνέπειες. Πρόκειται για δύο κανονισμούς που δεν ξέρω πώς μπορούμε να τις αλλάξουμε. Το θέμα της νομικής βάσης του 2007 και 2009 είναι αυτά τα δύο κείμενα. Αλλά επαναλαμβάνω, οι πολιτικές συνέπειες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Η πρόταση της Επιτροπής στο άρθρο 4, παραδείγματος χάρη, που αναφέρεται σε σημεία γνωρίζουμε σήμερα ποια μπορεί να είναι η συγκεκριμένη ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Καταλαβαίνετε ότι εδώ άτομα που δεν έχουν παραδείγματος χάρη την ε, ευρωπαϊκή η ηθαγένεια δεν θα συνυπολογίζονται σε αυτές τις ε, στατιστικές. Οι αποφάσεις λοιπόν θα ήταν πολύ πιο εύκολο να ληφθούν για κράτη-μέλη τα οποία παραδείγματο χάρη έχουν πάρα πολλούς μετανάστες. Στο άρθρο 2, 3, 4, Θεωρώ ότι τα δημογραφικά στοιχεία και οι προτάσεις για τις στατιστικές θα πρέπει να επανεξεταστούν. Επίσης η πρόταση για τους 12 μήνες, δηλαδή η χώρα υποδοχής πρέπει να ασχοληθεί με αυτούς τους ε, μετανάστες. Ξέρουμε όμως σήμερα ότι πολλοί επιστρέφουν στις χώρες τους, άλλοι όχι και άλλοι το κάνουν μετά τους 12 μήνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η μετανάστευση προς την Δυτική Ευρώπη είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί. Τώρα, εγώ έχω κάνει κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις και θα υποστήριζα ότι εδώ θα πρέπει να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στο κείμενο της Επιτροπής δεν λαμβάνονται με σοβαρό τρόπο υπόψη αυτά που μέχρι τώρα έχουμε πει. Θεωρώ ότι σε επίπεδο περιφερειών είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να καθορίσει τις στατιστικές. Υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες ξεπερνούν πολλές φορές τις διοικητικές ενότητες. Επίσης η έννοια του μόνιμου κατοίκου, είτε του προσωρινού κατοίκου. Εγώ εδώ θα ήθελα να καθοριστεί σε μία πενταετία και ο χαρακτηρισμός τη μου κατοίκου να είναι μετά τα πέντε χρόνια. Αυτά τα πέντε χρόνια για μένα είναι πραγματικά μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά, πεδίο αναφορά ιδιαίτερα για αυτού που ασχολούνται και με τα δημοσιονομικά θέματα. Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση του Άντριου Νταφ, όπως ξέρετε, επειδή είχε σαν θέμα πολύ ευαίσθητα, πολύ λεπτά ε, θέματα, έχει σταματήσει έχει βγει από το προσκήνιο και βεβαίως καταλαβαίνω τα επιχειρήματα αυτών που ασχολούνται με την δημογραφία και με τις στατιστικές. Εδώ υπάρχουν και αρμόδιες αρχές ε, στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών που έχουν ήδη δημοσιεύσει απόψεις και εκθέσεις, αλλά πολύ φοβάμαι ότι εδώ κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε πάρα πολύ σημαντικές ε, επαναλαμβάνω, ε, αρνητικές επιπτώσεις, σοβαρές πολιτικές επιπτώσεις. Περιμένω την υποστήριξή σας, περιμένω τις προτάσεις σας, καθότι θεωρώ ότι είναι αδύνατον να προχωρήσει αυτή η έκθεση της Επιτροπής ως έχει. Ε, Κυρία Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να δεχτώ την πρόταση διότι πράγματι χρειαζόμαστε μια, ένα κοινό πλαίσιο για να διαθέτουμε ακριβή στατιστικά στοιχεία πλήρη και συγκρίσιμα. Μέχρι τώρα τα στοιχεία συλλέγονταν επί εθελοντικής βάσης και αυτό είναι, ήταν πρόβλημα διότι τότε δεν είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία μιας χώρας μέλους με τα στοιχεία μιας άλλης. Αυτή η έλλειψη λοιπόν κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου σε εποχή όπου χρειαζόμαστε τέτοια στοιχεία γιατί αντιμετωπίζουμε δημογραφικές προκλήσεις είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρξει κοινή νομοθεσία σε ενωσιακό επίπεδο δεν υπήρχαν ούτε κοινέ έννοιε ούτε κοινοί ορισμοί μέχρι τώρα. Πρέπει να εναρμονιστούν όλα αυτά και τα χαρακτηριστικά, τα κριτήρια της συλλογή των στοιχείων, να έχουμε πολύ ψηλού επίπεδου κριτήρια και να έχουμε συγκρίσιμα αποτελέσματα και φυσικά να έχουμε συγκεκριμένες πηγές των στοιχείων και μεθόδους υπολογισμού που να είναι αξιόπιστες και να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν όλες οι χώρες μέλη. Τώρα νομίζω ότι ο στόχος της έκθεσης αυτής είναι επίσης πολύ σημαντικός γιατί θα καταλήξει σε αναρμόνιση των στοιχείων για ένα πολύ σημαντικό θέμα, τις δημογραφικές διακυμάνσεις. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει το ίδιο πλαίσιο αναφοράς για όλους και βέβαια τα πράγματα θα διευκολυνθούν αν μπορέσουμε να έχουμε αξιόπιστα στοιχεία για τις γεννήσεις, τους θανάτους, το προσδόκιμο ζωής, τις και ροές κτλ. Έχουμε όμως μερικές αμφιβολίες όπως την αναγκαιότητα να διαγραφούν μερικές από αυτές τις συστάσεις γιατί άκουσα άλλους να μιλούν για περιφέρειες όπου φαίνεται ότι υπάρχουν πολιτικές διαφορές ότι πολιτικός είναι, η πολιτική είναι η βάση της πρότασης διαγραφής μερικών από αυτές τις παραγράφους. Θα το μελετήσουμε, γιατί φοβόμαστε ότι η ταξινόμηση σε παραμένει πολύ σημαντική και η αλλαγή της θα ήταν κάτι ιδιαίτερα δύσκολο εφόσον θέλουμε να υπάρξει και περιφερειακή ολοκλήρωση και συνδυασμός των στοιχείων. Πρέπει να μας εξηγήσουν όσοι διαφωνούν τι εννοούν. Δεν μπορώ να σας πω από τώρα αν θεχόμαστε τις διαγραφές αυτές που ζητήθηκαν. Θα το μελετήσουμε όμως και ο εισηγητής μίλησε και για το αίσθημα του ανήκειν εθνικός. Τι θα πει αυτό το ανήκειν. Εδώ γράφει ότι πρόκειται για μία εθνοπολιτιστική ταύτιση με κριτήρια τη γλώσσα ή τον πολιτισμό. Εμείς αναρωτιόμαστε για ποια γενιά μιλάμε πόσες γενιές εφαρμόζεται αυτό το κριτήριο. Δεν είναι φανερό μέχρι πού θέλουμε να τα εφαρμόζουμε. Ούτε έχει νόημα να χωρίζουμε τα στοιχεία με βάση τέτοια κριτήρια ε, εθνότητας, γλώσσας κλπ. Ο εισηγητής μας λέει απ' την άλλη ότι αντί να είναι λίγη διορία τα μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου προτιμάει 0 η ώρα 1η Ιανουαρίου. Δεν την καταλαβαίνω τη διαφορά. Επίσης δεν είδαμε και πολύ μεγάλη συνένεση. Απλώς ότι χρειάζονται στατιστικά στοιχεία που πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη, συνεπή και συγκρίσιμα. Νομίζουμε ότι χρειάζεται εδώ νομοθεσία και θα επανέλθουμε με τροπολογίες και συστάσεις μέχρι τις 23 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάνερ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον συγγετή για αυτό το εξαιρετικό έργο. Θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντική η έκθεση αυτή, βέβαια είναι τεχνική, αλλά όπως ε, διαπιστώσαμε χρειαζόμαστε σήμερα ένα κοινό πλαίσιο. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα στοιχεία σε σχέση με τις ε, στατιστικές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κανονισμός αυτός ε, για τη δημογραφία να μπορεί να είναι ξεκάθαρος, ε, γιατί πολλές φορές διαφέρουν τα συστήματα μεταξύ των κρατών μελών, κυρίως ό,τι αφορά τα μητρώα. Με επιτρέπετε να αναφέρω κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν επιμέρους άρθρα. Θα έπρεπε να τροποποιηθεί το άρθρο 3, όπου αναφερόμαστε στον τόπο κατοικίας ε, και στην ε, πολιτογράφηση. Θα πρέπει να καταστήσουμε πιο ισορροπημένο τον κανονισμό για να υπάρχει καλύτερο συντονισμός κατόπιν. Τα κράτη-μέλη όταν εκπονούν τις στατιστικές θα πρέπει να είναι σε θέση να, λαμβάνουν υπόψη όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο Έχουμε την αναφορά του επίσημου τόπου κατοικίας, αλλά θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η έννοια αυτή ερμηνεύεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Στο άρθρο 4 έχουμε επίσης ε, τη μετακίνηση για συγκεκριμένο σκοπό. Πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό και θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται με την επίσημη κατοικία, με τον επίσημο τόπο κατοικίας. θα έπρεπε να έχουμε εδώ τον ίδιο ορισμό με αυτό που χρησιμοποιείται στο άρθρο 2. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε σαφέστατους ορισμούς. Όλοι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα τεχνικά στοιχεία, αλλά είναι σημαντικό να είμαστε πάρα πολύ ακριβείς και αυτό θα το πράξουμε μέσω της κατάθεσης τροπολογιών. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Όρη. Και κατόπιν, αφού ζητά το λόγο, θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο των Κομισιών και θα ολοκληρώσουμε τη γενική συζήτηση. Παρακαλώ, κύριε Σόρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να προσθέσω και εγώ δύο λόγια για το θέμα αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω την προσοχή σας σε αυτά που προτείνει ο εισηγητής. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να συζητάμε για το όσο αυτός προτείνει. Αυτό φυσικά δεν είναι καινοτομία. Έχουμε πολλές φορές ε, τεχνικές γνωμοδοτήσεις, ε, όμως ε, ξέρετε παρά όλο που είναι τεχνικές, οι πολιτικές επιπτώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Δεν συμβαίνει αυτό πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι εμπειρογνώμονες στις στατιστικές προτείνουν το εξής. Αυτό που προτείνουν είναι να μπορούν να συγκρίνουν τις στατιστικές. Όμως είναι δική μας ευθύνη, δικό μας καθήκον να δούμε και την πολιτική επίπτωση, της πολιτικές πτυχές αυτής της έκθεσης να τα βάλουμε στη ζυγαριά και να δούμε τι πολιτικά προβλήματα, επαναλαμβάνω, μπορεί να προκαλέσει. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ποια μέθοδο εργασίας θα ακολουθήσουμε, πώς δημιουργούνται αυτά τα στατιστικά στοιχεία, βάσει ποιας μεθόδου, ποιας μεθοδολογίας και βεβαίως να δούμε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι εκλογικό αποτέλεσμα θα προκαλέσουν. Καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάω μόνο για τις εθνικές είτε τοπικές εκλογές, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο συμβουλίου. Επαναλαμβάνω, ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Η κινητικότητα λοιπόν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι που βεβαίως θέλουμε να το ενισχύσουμε, να το προωθήσουμε. Υπάρχουν πολλά μέτρα που θα μας οδηγήσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά η διάσταση αυτή θα πρέπει να σταθμιστεί και επαναλαμβάνω αυτή η φαινομενικά τεχνική ρύθμιση ε, έχει, και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, πολιτικές επιπτώσεις. Δεν βιαζόμαστε, χρόνο έχουμε, θα πρέπει να το σκεφτούν και οι άλλες πολιτικές ομάδες και με τους κοιόδης εισηγητές ε, θα συναντηθούμε και θα δούμε πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα για μένα. Έχει δίκιο ο κύριος Σόγκαρ. Πρόκειται για μια τεχνική έκθεση, η οποία όμως στο μέλλον θα έχει και θα προκαλέσει σοβαρά πολιτικά προβλήματα. Οι εμπειρογνώμονες έχουν κάνει εδώ μια πολύ ασφαλμένη παρουσίαση και είναι δική μας αποστολή να δούμε και να εξετάσουμε και τις πολιτικές επιπτώσεις. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριο Μπερντό, ο οποίο είναι διευθυντή της Eurostat. Παρακαλώ. Μικρόφωνο παρακαλούμε για τον ομιλητή. Excuse me. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή και ευχαριστώ και τους ε, βουλευτέ για τα σχόλια. Νομίζω ότι υπάρχει κοινή συμφωνία ότι χρειάζεται κοινή νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις δημογραφικές στατιστικές και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την Κομισιόν. Όπως σας είπα, αυτός ο σημαντικός τομέας των στατιστικών σήμερα καλύπτεται με συμφωνίες κυρίων τα ευρωπαϊκά όργανα, το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν χρειάζονται πληροφορίες υψηλής σημασίας ε, για σημαντικά γεγονότα. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για διοικητικούς σκοπούς και ιδίως για το σύστημα της ειδικής πλειοψηφία στο Συμβούλιο και για την κατανομή των διαφορετικών ταμείων. Επίση υπάρχουν πάρα πολλοί παρανομαστές στα στοιχεία που παράγονται. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικά για την παρακολούθηση της στρατηγικής ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να έχουμε νομοθεσία προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι προφανές επίσης ότι η αυστηρή συγκρισιμότητα των πληροφοριών πρέπει να επιτευχθεί για ε, τους σκοπούς της ε, ψηφορία ειδική πλειοψηφία. Η Κομισιόν επιμένει ε, στο να υπάρχει ένα αυστηρό ορισμό τη κατοικία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να υπάρχουν εναρμονισμένα και συγκρίσιμα κριτήρια. Σύμφωνα με τις διεθνείς συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών ε, ή ε, ορισμός της συνήθους κατοικίας ε, πρέπει να βασίζεται σε μία περίοδο αναφοράς 12 μηνών. Αυτό είναι ο ορισμός των Ηνωμένων Εθνών. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να παραμένουμε σε ορισμούς που έχουν συμφωνηθεί διεθνώς για να αυξήσουμε την αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων, γιατί αυτό αυξάνει και την αξιοπιστία της όλης διαδικασίας. Αυτό πράξαμε πριν 10 χρόνια περίπου όταν ε, συστήσαμε τους δείκτες ε, για την ε, Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, δηλαδή τους δείκτες του Μάστρικτ. Είδαμε ποιοι είναι οι συμπεφωνημένοι δείκτες και χρησιμοποιήσαμε τους δείκτες αυτούς για να ορίσουμε το χρέος και το έλλειμμα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το να μείνουμε σε αυτές τις διεθνώς συμπεφωνημένες έννοιες είναι κάτι που επιφέρει αξιοπιστία στην όλη διαδικασία και το ίδιο ισχύει και για την ταξινόμηση των ΝΑΤΣ που αναφέρθηκε. Επίσης, ε, το όλο σύνολο των ε, στατιστικών για τον πληθυσμό βασίζεται στο δύο έχουμε ε, τις χάρη στατιστικές για τη μετανάστευση, στατιστικές απογραφών που χρησιμοποιούνται οι δύο ορισμοί. Επίσης πρέπει να λάβετε υπόψη ότι οποιαδήποτε παρέκκληση από αυτές τις συγκεκριμένε ταξινομήσεις ε, θα σημαίνει πρόσθετη προσπάθεια στις χώρες ε, και αύξηση ε, του άχθους και θα χρειαζόταν πιο συχνή χρήση των εκτιμήσεων και ο πιθανό, θα υπήρχε πιθανός αντίκτυπος στην ποιότητα των αριθμητικών στοιχείων. Θέλουμε λοιπόν εμείς ε, να έχουμε αυστηρή στοιχεία και για την ε, ψηφοφορία δικής πλειοψηφίας αλλά και για άλλους ε, σκοπούς, για κατανομές κονδυλίων και τα λοιπά. Οι χώρες μπορούν να χρησιμοποιούν τον όρο της συνήθως κατοικίας, αλλά αν δεν μπορούν θα δώσουμε κάποια ευελιξία για αυτές τις λεπτομέρειες. Και για να κλείσω, να σας πω ότι θα συμπληρωθεί αυτός ο κανονισμός από εφαρμοστικούς κανονισμούς της Κομισιόν, όπου θα έχουμε και όλα τα στοιχεία, τα τεχνικά που έχουν συμφωνηθεί και έχουν συζητηθεί σε τεχνικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, εισηγητής. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις διάφορες ερωτήσεις που ακούστηκαν. 31 Δεκεμβρίου ή 1η Ιανουαρίου. Στα έγγραφα που γνωρίζω, που είδα, πάντα υπάρχει η 1η Ιανουαρίου. Πάντα. Είναι τεχνικό ίσως το θέμα. Αλλά δεν έχω δει στη ζωή μου πουθενά να αναγράφεται η 31η Δεκεμβρίου σαν ημερομηνία. Τώρα, η υπηκότητα. Αν ήξερε η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, τα προβλήματα που θα είχαν αντιμετωπίσει αν όλοι αυτοί οι μουσουλμάνοι δεν είχαν ενσωματωθεί, αν το γνώριζαν εκ των προτέρων, θα είχαν ε, κάνει μια τελείως διαφορετική πολιτική. Τα στοιχεία, τα στατιστικά είναι πολύ σημαντικά, αλλά ακόμα πιο σημαντικά είναι ε, να αντιμετωπίσει κανείς τις επιπτώσεις αυτών των αριθμών. Εγώ αυτό που θέλω εδώ να πω είναι ότι είναι απαραίτητη η εναρμόνιση. Συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το είπα και αυτό αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι, αν θέλετε, κάτι που εξαρτάται από τις ε, αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Και τίποτα δεν μας υποχρεώνει εδώ να υιοθετήσουμε ακριβώς τις ίδιες προτάσεις. Σήμερα βλέπετε ότι παίζουμε με τους αριθμούς και αυτό είναι αντίθετο με το πνεύμα της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πολλοί υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζουν εδώ, στο Βέλγιο. Πολλοί διερμηνείς, πολλοί ευρωυπάλληλοι ζουν στο Βέλγιο εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχουν διάφοροι αριθμοί. Περίπου 600.000 εργάζονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση και περίπου 400.000 μετανάστες. Καταλαβαίνετε ότι εδώ οι αριθμοί δεν λένε πολλά και το ίδιο θα έλεγα και για την Κύπρο. Στην Κύπρο παραδείγματος χάρη, όπως ξέρετε υπάρχουν διάφοροι αριθμοί. Το ίδιο θα έλεγα και για την Ρουμανία. Για τη Ρουμανία οι αριθμοί αυτών που εγκαταλείπουν την χώρα μας είναι κάτι που δεν μπορούσαμε αρχικά να το υπολογίσουμε. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικές, σοβαρές πολιτικές συνέπειες. Αυτό που θα ήθελα να πω. Και υπάρχουν κράτη-μέλη που πρέπει να μπορούν να υπολογίσουν, να συνυπολογίσουν αυτές τις πολιτικές συνέπειες. Γιατί μιλήσαμε για την 12 παραμονή και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το θέμα της διάρκειας. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που θέλω να πω πίσω από όλα αυτά τα σχόλια είναι ότι πίσω από μια φαινομενικά τεχνική πρόταση υπάρχουν σοβαρές πολιτικές συνέπειες, γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ναι. Σαν νομοθετική αρχή βρισκόμαστε συχνά αντιμέτωποι με κάτι που φαινομενικά φαίνεται τεχνικό, πίσω όμως από το τεχνικό υπάρχει το πολιτικό. Γι' αυτό και δεν πρέπει πάντα να αφήνουμε τον έλεγχο στους εμπειρογνώμονες. Χρειαζόμαστε τους εμπειρογνώμονες, δεν αρνούμε την χρησιμότητά τους, αλλά οι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από εμά. Αγαπητέ συνάδελφοι, 23 Οκτωβρίου στις 12 είναι η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών και θα εξετάσουμε στις 28 Νοεμβρίου τις τροπολογίες αυτές. Θα ψηφίσουμε στις 29 Νοεμβρίου. Νομίζω ότι έληξε η συνεδρίαση. Ζητώ από τους συντονιστές να παραμείνουν όμως στην αίθουσα για λίγα λεπτά και θα ξανασυναντηθούμε εδώ το απόγευμα στις 3.